Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε αγαπητοί συνάδελφοι την απογευματινή μα συνεδρίαση. Θα ήθελα να εξηγήσω στους καλεσμένους μας ότι συνήθως ξεκινάμε στις 3 την απογευματινή μας συνεδρίαση. Αλλά σήμερα δεδομένες της ημερήσιας διάταξης και των πολλών σημείων που έχουμε να διεκπαιρεώσουμε ε, αρχίζουμε μισή ώρα νωρίτερα. Γι' αυτό ίσως δεν έχουμε τόσο πολλούς συναδέλφους. Και επειδή πολλοί έχουν ακόμη στο μυαλό τους τη τρεις, γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγο στην έναρξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Ζωάο Φιγκερέιντο, που είναι μέλος του πρώτου σώματος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και θα μας παρουσιάσει την έκθεση που εκπώνησε το Ελεκτικό Συνέδριο επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωρική πολιτική μετά το 2020. Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 7 Νοεμβρίου. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020 θα έχει τεράστια σημασία και για τη δική μας Επιτροπή, για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τους γεωργούς φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα η γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντική και για μας, γιατί το ελεκτικό συνέδριο πραγματοποιεί μια ανεξάρτητη υψηλό επίπεδο αξιολόγηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί συζητήσαμε δύο νομοθετικές προτάσεις που αφορούν αυτή τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και σίγουρα εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου. Και θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα της έκθεσής σας. Πάντως είναι πολύ αγαστή συνεργασία που έχουμε με το ελεκτικό συνέδριο γιατί ε, είναι αμοιβαίως επωφέλης αυτή η συνεργασία. Ασχολούμαστε λοιπόν με την πραγματοποίηση της, με την σύνταξη, χάραξη, εφαρμογή και εποπτεία της κινηζιωρικής πολιτικής. Και φροντίζουμε όλοι να είναι στο δυνατό πιο άρτια γίνεται και ιδιαίτερη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ μετά το 2020. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Φιλ Χόγκαν, που ήρθε για να συζητήσουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που θα μας παρουσιάσει ο κύριος Φιγκερέντο και θα λάβει μετά το ελεκτικό συνέδριο το λόγο για να μας σχολιάσει τη μελέτη αυτή. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Φιγκερέντο να μας κάνει την παρουσίαση μέσα σε ένα τέταρτο αν γίνεται. Θα το είμαστε ευγνώμονες αν τηρούσε αυτό το χρονικό περιθώριο και μετά θα ακούσουμε τον Επίτροπο Χόγκαν. Και καλωσορίζω θερμά και το επιτελείο σας. Μπορούμε λοιπόν να ακούσουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου πρώτα. Κύριε Φιγκερέντο, έχετε το λόγο. Thank you, thank Chair. Uh, first all, I would like to thank... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που στείλατε στο ελεκτικό συνέδριο για να σας παρουσιάσω από πρώτο χέρι τη γνωμοδότησή μας, την έκθεσή μας για το την ΚΑΠ μετά το 2020 και μάλιστα ε, έχουμε υποχρέωση να λαμβάνουμε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά δεν είναι μόνο υποχρέωση και καθήκον μας να παίρνουμε μέρος στη συζήτηση αυτή, είναι και ευχαρίστηση για μας ε, να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε επίγνωση της σημασίας που θα έχουν οι νέοι κανονισμοί για την κοινή γεωρική πολιτική. Και το γνωρίζουμε αυτό γιατί η κοινή γεωρική πολιτική αντιπροσωπεύει ένα τεράστιο τμήμα του ενωσιακού προπολογισμού. Οπότε είναι υποχρέωση καθήκον του ελεκτικού συνεδρίου να κατανοήσει πλήρως και αυτό επιχείρημα να κάνουμε τα σχετικά με τους κανονισμούς για τη νέα ΚΑΠ. Μάλιστα θα χρησιμοποιήσω κάποιες διαφάνειες, ένα PowerPoint για να διανθίσω την παρουσίασή μου. Καταρχήν θα σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο δεν είναι πολιτικό σώμα. Εσείς είστε οι πολιτικοί θύνοντες για τη χάραξη πολιτικής. Οπότε θα σας παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία που διέπουν τις γνωμοδοτήσεις μας. Καταρχήν, το πρώτο θεμέλιο της έκθεσης είναι οι γενικές αρχές των δημοσίων πολιτικών. Θέλουμε μια σωστή ε, σωστό ορισμό των ε, δημοσίων αναγκών. Να δούμε αν οι ανάγκες προσδιορίζονται επαρκώς και αν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό είναι ουσιώδη στοιχείο μιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Επίσης, ε, διερευνούμε κατά πόσο προσδιορίζονται σωστά οι στόχοι αυτής της δημόσιας πολιτικής που είναι κοινή γεωρική πολιτική. Θέλουμε να δούμε αν τα επιμέρους στοιχεία, οι συνιστώσεις της πολιτικής προσδιορίζονται σωστά. Οι διαδικασίες της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής είναι άρτιες. τα αποτελέσματα έχουν ε, ε, καλό σχεδιασμό και καλές συνέπειες. Και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει πολύ είναι αν οι μηχανισμοί της λογοδοσίας που προβλέπουν νομοθετικές προτάσεις είναι σωστοί και ευθυγραμμίζονται με τις γενικές αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αυτά λοιπόν είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που διέπουν την έκθεσή μας, την γνωμοδότησή μας. Άλλο σημαντικό θέμα θεμελιώδης είναι η συνοχή και η συνέπεια της πολιτικής, η συγκρότησή της. Ε, θα διερευνήσουμε κατά πόσο η μεταρρυθμισμένη κοινή γεωρική πολιτική είναι συνεκτική και συνάδει και με τις υπόλοιπε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στηρίζουμε τις γνωμοδοτήσεις μας και σε προηγούμενες ε, ε, εκθέσει και μελέτες μας και σε προηγούμενα πόρισματά μας. Θα δούμε λοιπόν τι πορίσματα είχαμε εκδώσει στο παρελθόν για τους επιμέρους μηχανισμούς και πολιτικές και θα σας υπενθυμίσω τις προηγούμενες μελέτες ε, και γνωμοδοτήσεις μας. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι καταρτήσαμε την γνωμοδότησή μας βάσει της συνθήκης και μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο της γνωμοδότησής μας. Χωρίστε σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα κάνει έναν ορισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής, που είναι μια γεωργική πολιτική και μετά θα σας δώσω τη γνώμη μας για το νέο μοντέλο παρουσίαση αποτελεσμάτων, το delivery model. Σε ό,τι αφορά την, τον ορισμό της CAP. τα βασικά μας μηνύματα είναι τα εξής. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι κατά τη γνώμη μας δεν είναι σαφές ε, ή εμφανές ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη μεταρρυθμισμένη ΚΑΠ. Δεν λέμε ότι δεν έχουν γίνει μελέτες, ότι δεν υπάρχουν σενάρια, γιατί και μελέτες υπάρχουν και πολλά σενάρια. Αλλά δεν αφήνουν αυτά να διαγραφεί με σαφήνεια ένα μακροπρόθεσμο όραμα της ΚΑΠ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι σαφές τουλάχιστον. Ούτε για την ΚΑΠ ένα μακροπρόθεσμο όραμα, ούτε για τους μηχανισμούς της. Αυτό είναι το πρώτο μας μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι δεν έχουμε βρει ε, στιβαρά οικονομικά πιστήρια ή ενδείξεις για τους βασικούς μηχανισμούς της ΚΑΠ. Και κυρίως δεν βρίσκουμε ε, αρκετά πιστήρια, ε, στιβαρές ενδείξεις για το μεγάλο ρόλο των άμεσων ενισχύσεων. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Στοιχεία υπάρχουν και πολλά μάλιστα. Υπάρχουν και πολλοί επιχειρήματα αλλά δεν βλέπουμε ισχυρά πιστήρια υπέρ της διατήρησης αυτών των μηχανισμών, όλων των μηχανισμών της ΚΑΠ. Γιατί η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή γεωρική πολιτική, ουσιαστικά συνεχίζει τους μηχανισμούς της παλιάς ΚΑΠ. Τρίτο μήνυμα. Κατά τη γνώμη μας, οι περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι σημαντικές και αναφυσβήτητες στο μέλλον θα εξαρτηθούν από τις επιλογές των κρατών μελών και από τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εθνικές επιλογές στα περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα. Δεν ξέρουμε με τι κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις στο μέλλον. Και θεωρούμε ότι ε, μία συνεισφορά της ΚΑΠ σε επίπεδο 40% για την υλοποίηση Τη κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική, μια τόσο υψηλή συνεισφορά της ΚΑΠ τη τάξη του 40% για τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους είναι ουτοπική κατά τη γνώμη μας, δεν είναι καθόλου ρεαλιστική. Και αυτό το πόρισμα το στηρίζουμε σε προηγούμενες μελέτες και γνωμοδοτήσεις μας. Τέταρτο συμπέρασμα. Οι συντελεστές χρηματοδότησης δεν αντικατοπτρίζουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία είναι μια κρίσιμη πτυχή της νέας πολιτικής. Και δεν βλέπουμε έναν ξεκάθαρο σύνδεσμο μεταξύ των συντελεστών σε χρηματοδότησης και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Τέλος. Υπάρχει και ένα νέο στοιχείο στην ΚΑΠ ένα καινοτόμο στοιχείο σε σχέση με την παρούσα ΚΑΠ. Το νέο αυτό στοιχείο είναι τα ανώτατα όρια των πληρωμών, το κάπινγκ. Θεωρούμε ότι τα ανώφυλα πληρωμών στις μεγάλες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα είναι περιορισμένα αν το κόστος της εργασίας αμοιβόμενης και μη αποκλείεται από το ανώτατο όριο από την άλλη πλευρά, αν λάβουμε υπόψη το εργασιακό κόστο, τη αμοιβόμενη και μη εργασίας, αυτό θα αποδυναμώσει τα αποτελέσματα της θέσπισης ανωτά των όριων του κάπινγκ. Αυτά είναι τα βασικά μας μηνύματα ως προς τον ορισμό της κοινή γεωργική πολιτικής. Τώρα, ποια είναι η γνώμη μας για το νέο μοντέλο παροχής αποτελεσμάτων, το delivery model της ΚΑΠ. παρόλο που ως προς την πολιτική, την κοινή γεωργική πολιτική δεν θα αλλάξουν πολλά, γιατί οι βασικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Η συμμετοχή της στον ενωσιακό προϋπολογισμό επίση είναι παρόμοια. Αλλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές ως προς το νέο μοντέλο που χρησιμοποιεί η ΚΑΠ, που είναι το μοντέλο που βασίζεται στα αποτελέσματα. Είναι το delivery model και στηρίζεται σε τέσσερις ε, έννοιες. Την επικουρικότητα, την επίδοση, την απλούστευση και τη λογοδοσία. Μια και δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί μόνο πέντε λεπτά μου έχουν απομείνει, θα σταθώ μόνο σε δύο έννοιες, στις επιδόσεις και στην λογοδοσία. Τι γίνεται λοιπόν με τις επιδόσεις και τη λογοδοσία στους νέους κανονισμούς για την ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά την επίδοση, τις επιδόσεις. Κατά τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου, γίνεται μια σωστή κίνηση προς ένα σύστημα που θα εδράζεται στις επιδόσεις, ε, στα αποτελέσματα. Αυτή η κίνηση είναι καλή. Θεωρούμε όμως ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος βάση επιδόσεων. Καλή μένει προσπάθεια, αλλά λείπουν βασικά στοιχεία από ένα σύστημα που βασίζεται στις επιδόσεις. Γιατί θεωρούμε ότι λείπουν τα στοιχεία. Γιατί είναι βασικά στοιχεία όπως σαφής, συγκεκριμένη και ποσοτικοποιημένη ευρωπαϊκή στόχοι για να καταμετρηθούν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα. Γιατί αν θέλουμε επιδόσεις, χρειαζόμαστε προηγουμένως στόχους. Και αν θέλουμε να κρίνουμε αν, έχουν, αν είναι καλέ επιδόσεις, θα πρέπει να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους. Γιατί χωρίς στόχους, πώς θα καταμετρήσουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με τι θα καταμετρήσουμε τα αποτελέσματα. Ένα άλλο στοιχείο που λείπει είναι σαφή σύνδεσμο, σαφή αλληλεπίδραση μεταξύ των μέτρων και των στόχων, γιατί ούτε και εκεί υπάρχει σαφήνεια. Επίσης, μας λείπει μία πλήρης δέσμη δικτών που αφορούν την παραγωγή, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο. Χρειαζόμαστε μία δέσμη δικτών, ένα σύνολο δικτών για τα αποτελέσματα, την παραγωγή και τις συνέπειες. Και μάλιστα στα παραρτήματα λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις για να καταλήξουμε σε ένα άρτιο σύστημα, άρτιο σύνολο δικτών. Αυτά ως προς τις επιδόσεις. Τώρα, ποια είναι η γνώμη μας για τη λογοδοσία. Σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία, άποψη μας είναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για το ελεγκτικό συνέδριο και φαντάζομαι θα είναι πολύ σημαντικό και για το Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι η πρόταση οδηγεί σε ένα αποδυναμωμένο πλαίσιο λογοδοσίας. Και γιατί ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Γιατί λέγοντας απλώς ότι είναι θετικό στοιχείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα μπορεί να πιστοποιεί την εγκυρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των λογαριασμών. Ως προς αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι μηχανισμοί για τους λογαριασμούς είναι σωστοί στους νέους κανονισμούς. Θεωρούμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει την ικανότητα να δηλώσει για το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών να δηλώσει κατά πόσο οι πληρωμές που έγιναν στους τελικούς δικαιούχους πληρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ε, εκείνα τα τμήματα των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Με τους λογαριασμούς δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την διαπίστωση αν οι πληρωμές ε, και τα, και τα στρατηγικά σχέδια πληρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ο Γενικός Δημοσιονομικός ε, Κανονισμός που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αναφέρει ότι οι λογαριασμοί θα πρέπει να συνοδεύονται από τη γνώμη ενός ανεξάρτητου ελεκτικού σώματος που θα ε, πιστοποιεί ότι οι δαπάνες ήταν νομότυπες και κανονικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στις δαπάνες της ΚΑΠ στο μέλλον θα έχουμε δύο διαφορετικά είδη δαπανών, δύο κατηγορίες δαπανών. Η μία κατηγορία αφορά τις δαπάνες που βρίσκονται εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Και έχουμε και τις δαπάνες που εμπίπτουν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Που, ε, μάλλον που είναι εκτός των στρατηγικών σχεδίων. Οι δαπάνες εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ είναι το 2%. Οι δαπάνες εντός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ είναι 98%. Στην πρώτη κατηγορία των δαπανών, το 2% δηλαδή, εκτός των στρατηγικών σχεδίων, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε κατά πόσο οι δαπάνες είναι νομότυπες και κανονικές. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τη δεύτερη όμως κατηγορία που αφορά το 98% των δαπανών της ΚΑΠ, εκεί διαπιστώνουμε ότι θα γίνει μία αξιολόγηση ως προς την υποβολή εκθέσεων για τις επιδόσεις και θα κριθεί αν είναι σωστή η υποβολή εκθέσεων, αν τα αποτελέσματα είναι σωστά. Εντάξει, αυτό είναι καλό και θετικό. Επίσης, στο μέλλον θα έχουμε μία αξιολόγηση των συστημάτων διακυβέρνησης. Δηλαδή, κατά πόσο τηρούνται ε, τα βασικά στοιχεία, τα, οι βασικές απαιτήσεις ένωσης από, τις, από τους φορείς διακυβέρνησης. Για το 98% των δαπανών δεν θα έχετε καμία επαλήθευση, κανέναν έλεγχο από ανεξάρτητο ελεκτικό φορέα για το κατά πόσο οι πληρωμές που έγιναν στους τελικούς ε, δικαιούχους πληρούν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δεν θα έχετε καμία τέτοια διαβεβαίωση με βάση το νέο σύστημα. Είναι σημαντικό αυτό για μας γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει συγκεκριμένους κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται από τους τελικούς δικαιούχους. Οπότε το Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου, το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να γνωρίζει κατά πόσο οι κανόνες που ενέκρινε τηρούνται στα κράτη-μέλη. Στο τελευταίο στάδιο των πληρωμών, των δαπανών. Και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει εξακρίβωση από ανεξάρτητο ελεκτικό φορέα για το κατά πόσο οι πληρωμές που έγιναν στους τελικούς δικαιούχους πληρούν την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία και ε, τα τμήματα των στρατηγικών σχεδίων που απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βέβαια, εσείς θα αποφασίσετε αν θέλετε ή όχι κάτι τέτοιο. Αν όμως δεν θέλετε να γίνουν τέτοιες επαληθεύσεις, τέτοιοι έλεγχοι. Θα ήθελα εγώ ως έλεγκτης και ως μέρος του ελεκτικού συνεδρίου να σας ρωτήσω, ε, τότε γιατί εγκρίνετε κανόνες για τους τελικούς δικαιούχους αν δεν πρόκειται να, τους, να ελέγξετε την εφαρμογή τους στο τελικό στάδιο. Προστίτωτε οι κανόνες αν δεν ελεγχθεί η εφαρμογή τους. Τέλος. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα διεθνές πρότυπο για τον έλεγχο. Εμείς ως ελεκτικό συνέδριο πληρούμε αυτό το πρότυπο. Φυσικά χρειάζονται διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου και υπάρχουν τέτοιες στους κανονισμούς. Επίσης χρειάζονται κάποιοι έλεγχοι, περαιτέρω έλεγχοι και ελεκτικές διαδικασίες και ε, δοκιμές των ελέγχων και ουσιαστικές διαδικασίες μαζί με δοκιμές λεπτομεριών και ουσιαστικές αναλυτικές διαδικασίες. Και δυστυχώς τέτοιες ε, ουσιαστικές διαδικασίες δεν έχουμε στους νέους κανονισμούς για την ΚΑΠ. Αυτό είναι πρόβλημα για μας σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία. Θέλουμε ουσιαστικές προ... διαδικασίες από ανεξάρτητους ελεκτικούς φορείς. Αυτό μέχρι στιγμής απαιτείται μόνο για το 2% των δαπανών, για, τον, για τις δαπάνες δηλαδή που εκπίπτουν, που βρίσκονται εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Και αυτό είναι το πρόβλημα που εντοπίζουμε σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία. Επίσης, από ένα μοντέλο που εδράζεται στη συμμόρφωση, μετακινούμαστε σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στα αποτελέσματα, στο delivery model. Τώρα, αυτή η καταστροφή έρει την ανάγκη για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των κανόνων που προβλέπουν οι κανονισμοί. Ε, κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι υπόλοιπε ε, συναλλαγές δεν θα ε, είναι πλέον πληρωμές τελικούς ε, δικαιούχους, αλλά μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε, πια δεν θα ελέγχονται οι, οι δαπάνες της ΚΑΠ εντός των κρατών μελών, παρά μόνο οι μεταφορές κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Αυτά, επειδή έχω εξαντλήσει το χρόνο μου, θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Φιγκερέιδο. Πραγματικά ήταν πολύ σαφής η παρουσίαση και τηρήσατε και το χρόνο σας. Ακούσαμε την γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα ακούσουμε τώρα και τον Επίτροπο Φιλ Χόγκαν για να μας πει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Φιγκερίδου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία δημοσία να τοποθετηθούμε σε σχέση με τη γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου και την πρόταση μας για την περίοδο μετά το 2020. Εξ αρχής σας λέω ότι πάντοτε είχαμε καλή επικοινωνία η ε, Επιτροπή σας και η Γενική μας Διεύθυνση. Βέβαια να δούμε αν αυτό θα συνεχίσει να ισχύει όταν ολοκληρώσω αυτό που έχω να σας πω. Πάντως χρειάζεται να σχολιάσουμε τα της γνωμοδότησης γιατί σε πολλά σημεία διαφωνώ. Πρώτα-πρώτα αισθάνομαι απογοήτευση γιατί μετά την ανακοίνωση που διέρευσε δεν είχα την ευκαιρία να μελετήσω τα, τα περιεχόμενα και το περιεχόμενο οπότε από την αρχή ήμουν αρνητικά προδιατεθειμένος και οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί που ξέρουμε τα θέματα, εκεί που έχουμε αρμοδιότητα και εμείς δεσμευτήκαμε να κάνουμε μια ανάλυση, ενδελεχή της γνωμοδότησης και γι' αυτό και θα σας μιλήσω. Εμείς απορρίπτουμε πολλά από αυτά τα συμπεράσματα που ακούσαμε και τα είπαμε και μπροστά στο Ελληνικό Συνέδριο, τα κοινοποίησαμε και σε εσά. Νομίζω ότι όλα αυτά οφείλονται σε παρερμηνίες, σε παρεξηγήσεις σε σχέση με τη θέση μας. Αυτό είναι λυπηρό. από αρχάς του 2017 έχουμε μία συνεννόηση, μία δέσμευση και από τον Ιανουάριο σε σχέση με το ελληνικό συνέδριο μια ολόκληρη μέρα περάσαμε με τον διευθυντή του ελληνικού συνεδρίου για κάποια ενημέρωση, για κάποια δεδομένα, ανάλυση, αξιολόγηση για τα θέματα της χάραξης πολιτικής. Πολλούς μήνες συνεργαστήκαμε ήταν ναι, η διαδρομή αυτή ανοιχτή και με διαφάνεια. Οπότε 16 δεκάτου ενεστώτος έτους απίφθηνα μια επιστολή στο συνέδριο και είπαμε τις θέσεις μας, είπαμε γιατί θέλουμε το καινούργιο delivery model για την ΚΑΠ, για επικουρικότητα, για επιδόσεις και είπαμε ότι αυτά θα μπορούσε να τα πάρει υπόψη το συνέδριο. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία ισχυρίζει το συνέδριο δεν είναι βάσιμα. Έχουμε ας με την μελλοντική αρχιτεκτονική, τους στόχους της ε, ΚΑΠ, το εισόδημα, τις άμεσες ε, ενισχύσεις, την ε, εξασφάλιση της προμήθειας των διατροφής, την προσφορά στο δημόσιο αγαθό. Κοιτάξτε, εμείς κατηγορηματικά διαφωνούμε με τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Είπαμε ότι θα πρέπει ρητός να καθορίζονται οι στόχοι για το κλίμα, τους φυσικούς πόρους και την βιοποικιλότητα. Εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα προαπαιτούμενα ε, και ιδίες όσον αφορά το νέο delivery model. Έχουμε τη νέα αρχιτεκτονική καλύπτει την ε, ενισχυμένη ερεσιμότητα για τον πρώτο πυλώνα. Πρασίνισμα για όλους τους και ε, καινούργια προγράμματα για τον πρώτο πυλώνα και τον δεύτερο πυλώνα. Οπότε είπαμε ότι καλύπτουμε 30% από το Ταμείο ε, Αγροτικής Ανάπτυξης. Και έχουμε μια σειρά άλλων παρεμβάσεων ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα, το περιβάλλον από πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Έχουμε και καινούργια στοιχεία, με μηχανισμούς, όπως ένα νέο άρθρο που λέμε τα κράτη-μέλη θα πρέπει έχουν σκοπό να συμβάλλουν περισσότερο όσον αφορά τους στόχους για περιβάλλον και κλίμα και να μην υπάρχει backsliding. Ε, ε, επίσης είπαμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους μπόνους που προβλέπονται ε, μιλάμε για την περίοδο 21 με 27 και έτσι συνδέουμε την ε, νομοθεσία για κλίμα και περιβάλλον με τα προγράμματα και την πολιτική για την γεωργία. Για τις άμεσες πληρωμές είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους γεωργούς, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Ε, για αυτό θα πρέπει να δούμε ε, το ότι το άρθρο 39 της συνθήκης τάσει τους σκοπούς της ΚΑΠ για βιωτικό επίπεδο των γεωργών, για το εισόδημα των γεωργών επίσης και το συνέδριο λέει ότι η αξιολόγηση είναι ανεπαρκής και ότι εμείς δεν έχουμε δώσει στεγανά στοιχεία, βάσιμα στοιχεία όσον αφορά αυτά τα μέτρα όπως οι άμεσες πληρωμές. Μα αυτό το μέτρο λέτε ότι θα πρέπει να καταργηθεί τελείως και λέτε ότι θα πρέπει να στηριζόμαστε σε στοιχεία, αλλά ενώ έχουμε για το εισόδημα στοιχεία, τα αγνοείτε. για την κατανομή του εισοδήματο, το επίπεδο, για τη συγκρισιμότητα με την υπόλοιπη οικονομία. Όλα αυτά είναι δημοσιοποιημένα. Κάναμε και αξιολόγηση επιπτώσεων και λέμε ακριβώς τις λεπτομέρειες που αφορούν το εισόδημα για τις εκμεταλλεύσεις και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για το πώς θα υπάρχει βιώσιμο εισόδημα, εξασφάλιση προμήθειας των διατροφής για να έχει μέλλον αυτή η υπόθεση και απευθύνομαι και στην Παγκοσμία Τράπεζα για την ΚΑΠ και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τον ρόλο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα στι άμεσες πληρωμές για απασχόληση, για ε, περιβάλλον όμως το συνεδρίο δεν το έκανε αυτό και αντί να δει τις επιπτώσεις Αντί να δει τις για το εισόδημα, ε, κοίταξε το εισόδημα εκτός κάπου, εκτό γεωργίας. Κοίταξε εθνική φορολογία, τα συνταξιοδοτικά, τα, κρατική πολιτική. Οπότε, εμείς θεωρήσαμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα λάβαμε υπόψη το 2017 μετά από διαβούλευση με το χάρτη πορεία στον οποίο καταλήξαμε. Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν σημαντικό και για θεσμικού λόγου το αφήσαμε την το τελικό κείμενο και ε, προσπαθήσαμε να είμαστε ε, συντονισμένοι επί τη συνθήκη. Τι λέει για την ΚΑΠ, ποιοι είναι οι στόχοι της ε, ΚΑΠ, λέει συνθήκη, όπως λέει για το βιωτικό επίπεδο των γεωργών, για την ε, διατροφική επάρκεια. Εμεί είμαστε ο εγγυητή των συμφύλακα των συνθήκων. Γι' αυτό και παραπέμπουμε στη μελέτη των επιπτώσεων, ε, παραπέμπουμε σε μελέτη που έγινε. Είπαμε ότι έχουμε 18% μείωση του εισοδήματο στην Ένωση και αυτό είναι χτύπημα για την οικονομική βιωσιμότητα της ε, υπαίθρου της γεωργίας. Έχουμε απερίμωση της ε, υπαίθρου και κίνδυνο για το περιβάλλον. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, έχουμε διάφορες εναλλακτικέ από αυτή τη μελέτη επιπτώσεων, έχουμε διάφορα μέσα πολιτικής, όπως προβλέπει η ΚΑΠ και είπαμε για ένα ελάχιστο επίπεδο αμέσων πληρωμών. Οπότε αυτού του είδους ε, η πολιτική στηρίζει το εισόδημα και από ό,τι φαίνεται η άμεση στήριξη στο μέλλον θα εξασφαλίσει τα, τα του κλίματος, το, τα του περιβάλλοντος, τα της υπαίθρου και έτσι φαίνεται το πόσο σημαντική είναι η ξεκάθαρη σχέση μεταξύ βιώσιμης γεωργίας και άμεσων πληρωμών. Για να δούμε τώρα ένα άλλο, δύο σημεία που θέλω να σχολιάσω. Όσον αφορά τόσο είπε το Συμβούλιο την Δευτέρα, είδαμε ότι για το νέο delivery model υπάρχει υποστήριξη. Η επιλεξιμότητα θα βασίζεται στο πόσο στεγανά είναι τα συστήματα διακυβέρνησης, τι γίνεται με την παραγωγή, να μην έχουμε ε, μέτρα για μεμονωμένους δικαιούχους. Σε αυτό το κείμενο λέμε ότι η παρέμβαση εξαρτάται από τη δέσμευση και συμμόρφωση των ε, δικαιούχων. Ε, αυτό είναι παραπλανητικό γιατί η νομική αρχιτεκτονική για το delivery model είναι ξεκάθαρη στην πρότασή μας. Το ίδιο ισχύει και για το κοινωτικό δίκαιο το οποίο θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές ε, διατάξεις. Το ίδιο ισχύει επίσης και τους οργανισμούς πιστοποίησης, τον έλεγχο του κατά πόσον τα εθνικά συστήματα λειτουργούν εύρυθμα και σας ε, διαβεβαίω ότι εμείς αυτό το ζήτημα της επιλεξιμότητας και της διακυβέρνησης το θέλουμε πάρα πολύ σομάρο Σοβαρό είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και να έχουμε καλές επιδόσεις και αυτό το αναγνωρίζει στην έκθεση το συνέδριο. Δηλαδή το τι διαχείριση θα γίνει ε, και έχουμε το 2,2% ως ποσοστό σφάλματος την τελευταία δεκαετία. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Όμως τώρα δεν το λέει αυτό το συνέδριο στην έκθεσή του. Δεν αναφέρεται στο πόσο πετυχημένο ε, είναι το σύστημα που έχουμε για τη διαχείριση των ε, ε, κοινωτικών πόρων για την γεωργία. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι έχουμε διαφορά στις απόψεις μας, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τα συμπεράσματα. Επίσης σας στείλαμε ένα παράρτημα αυτή τη εβδομάδα και εκεί διορθώνουμε, εκεί ξεκαθαρίζουμε κάποια από τα συμπεράσματά σας. Και παρακαλώ εσείς που είστε μέλη της Επιτροπής και νομοθέτες να προβληματιστείτε πάνω σε αυτά τα οποία λέμε. Μπράβο για το έργο που επιταλέσατε, για τις προτάσεις ε, αυτές και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα τα συζητήσουμε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι τον κοινό μας στόχο θα τον πετύχουμε. Να απλουστεύσουμε, να μεταρρυθμίσουμε την ΚΑΠ να έχουμε επιδόσεις, να έχουμε επίσης ε, επικουρικότητα. Οι στόχοι μας βασίζονται στα όσα τάση η ε, μελέτη ε, των επιπτώσεων. Και η αξιολόγησή μας που δεν έκανε το ελεγκτικό συνεδρίο, έχουμε εννέα στόχους που τα λέει η πρότασή μας. Εδώ βλέπετε τι αντικατοπτρίζεται από την κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή είναι συγκεκριμένη και εφικτή αυτή η στόχη για μια κοινή μας πολιτική. Και για κάθε στόχο διαλέξαμε κάποιους δείκτες για να υπάρξει παρακολούθηση των επιδόσεων και αξιολόγηση. Ε, θεωρούμε ότι αυτά είναι ρεαλιστικά και το σχέδιο κειμένου έχει επίσης ε, μία δέσμη των ε, δικτών για την παραγωγή, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε διαχείριση και αξιολόγηση των επιδόσεων. Καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο όλους τους στόχους και έτσι θα έχουμε και προγραμματισμό και αξιολόγηση. Οπότε με αυτούς τους δείκτες φτάσουμε τους στόχους αλλά και εφαρμόζουμε τον έλεγχο. Είναι αυτό η βάση της αξιολόγησης. Και όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια, τα κράτη-μέλη θα θέσουν με κάποιους, με κάποιους δείκτες, θα θέσουν κάποιους ε, στόχους για να πετύχουμε αυτά τα οποία πρέπει να πετύχει η ΚΑΠ. Άρα, σε επίπεδο κράτους μέλους θα βαδίσουμε επί τη βάση των επιδόσεων και όπως θέλουν τα κράτη-μέλη θα προσέξουμε τις επιπτώσεις πολιτικής και ε, την επίτευξη των στόχων. Να μην υπάρχει φόβος για τους ε, ελέγχους. Να υπάρχει λογική όσον αφορά την οικονομική διαχείριση της πολιτικής. Λυπάμαι που δεν συμφωνεί με αυτά το συνέδριο. Δεν προτείνουμε κάτι το οποίο να είναι κατά, να στρέφεται κατά του τελικού δικαίου με αυστηρούς κανόνες, με ελέγχους και δεν ωφελεί στην εξασφάλιση της ε, αυτάρκειας της προμήθειας ε, ειδών διατροφής. Είπαμε ότι δεν πετυχαίνει το παρόν σύστημα θα το αλλάξουμε. Άρα θα πρέπει να κρίνουν οι συνομοθέτες για το τι θα κάνουν. Θέλουν να το κάνουν, δεν θέλουν να το κάνουν, είναι δικαιωμά Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αφού ακούσαμε και τον Επίτροπο, θα δώσω το λόγο στις εισηγητριές μας και θα ακολουθεί η συζήτηση και με τους λοιπούς ευρωβουλευτές. Πρώτα η κυρία Ράς Γκαρσία που θα μας μιλήσει για τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια. Παρακαλώ κύριε Γκαρσία. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο και διάβασα την αιτιολογημένη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου πρώτα και μετά την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πιστεύω ότι η κριτική του ελεκτικού συνεδρίου το παρατραβάει, γιατί θέτεται σε αφιβολία το σύστημα άμεσων ενισχύσεων προς τους Γιώργους, που είναι η βασική υποστήριξη της κοινή γεωργικής πολιτικής για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματο. Ουσιαστικά δηλαδή επιτίθεστε κατά μέτωπο στο βασικό ε, στοιχείο της κοινή γεωργικής πολιτικής, που είναι το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου το στοιχείο όχι μόνο δεν θα πρέπει να επικρίνεται και θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά επιπλέον θα πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουμε την Ήπεθρο και τη Γεωργία, εκεί που, και κυρίως στις περιοχές που έχουμε μεγάλη δημογραφική πρόκληση ε, και πρόβλημα απερίμωσης και δεν μπορούμε ε, να ζητούμε από τη μια ασφαλή τρόφιμα και προσιτές τιμές όταν θα στερούμε από τους γεωργούς τη βασική υποστήριξη της κοινής γεωργικής πολιτικής. Γιατί μια τέτοια επίθεση αποβαίνει βάρος όχι μόνο των γεωργών, αλλά του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών που περιμένουν από τους γεωργούς ασφαλή και φθηνά τρόφιμα. Σε ό,τι αφορά τους ποσοτικοποιημένους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε και αυτό κατά τη γνώμη μου έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ διαφορετικές πραγματικότητες. Άλλο η Μεσογειακή Ευρώπη, άλλο η Λαπωνία. Έχουμε πολλά γεωγραφικά μήκη και πλάτη και πολύ διαφορετικά εδάφη, πολύ διαφορετικό κλίμα. Γι' αυτό περιμένουμε κάποιες ε, ε εκθέσεις, δάφο, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη αντίληψη για την κατάσταση κάθε χώρας. Γιατί Κάθε χώρα έχει διαφορετική πραγματικότητα, ιδιαιτερότητε, διαφορετικέ ανάγκε και γι' αυτό και η μεταχείριση θα πρέπει να είναι διαφορετική. Αν ακολουθήσουμε όμω τι δικέ σα οδηγίε του ελεκτικού συνεδρίου, θα οδηγηθούμε σε παταγώδη αποτυχία τη κοινή γεωρική πολιτική που ουσιαστικά θα τροφοδοτεί με επιχειρήματα του επικριτέ τη ΚΑΠ, που δεν είναι και λίγοι. Πιστεύω ότι στηριχθήκατε σε κάπως χολά επιχειρήματα. Φαίνεται ότι δεν ακούσατε καλά τις εξηγήσεις που δόθηκαν, γιατί οι διαβουλεύσεις ήταν δημόσιες. Σε όλες τις ε, συνεδριάσεις που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει προτάσεις της, η συζήτηση έγινε ξεκάθαρα και με σαφήνεια, μας το είπαν και τα λόμπι. Οι διαβουλεύσεις ήταν ευρύτατες. Όταν λοιπόν το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι το ο κανονισμός δεν προβλέπει βασικό σενάριο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, πώς είναι δυνατόν να έχουμε κοινή γραμμή εφόσον τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές πραγματικότητες. Αν δεν γίνει πρώτα μία εκτίμηση των, διαφορε... των ιδιαιτεροτήτων, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε στόχους, ούτε μέτρα, ούτε έλεγχο εφαρμογής των μέτρων. Είναι σαν να κάνουμε, εφαρμόζουμε προθύστερο σχήμα. Ούτε τις πληροφορίες λάβατε όντως υπόψη, ούτε αρκετή συνεργασία είχατε με τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τροφοδοτηθείτε με κατάλληλα στοιχεία. Ήταν κάπως εσπευσμένα τα απορίσματά σας. Και με τη συζήτηση των εκθέσεων βλέπουμε ότι διαπιστώ δημιουργείται μια σύγχυση και μια άγονη συζήτηση που δεν ε, τη διευκολύνεται καθόλου. Νομίζω ότι πρέπει καλύτερα να επικεντρωθούμε στα τεχνικά μέτρα. Σας ευχαριστώ. κύριε Σαντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βρισκόμαστε στην καρδιά της δημοκρατίας. Και σίγουρα η απόψη των συντηρητικών και των φιλελευθέρων δεν είναι ίδιες με αυτές των σοσιαλιστών. Αυτή είναι και η πεμπτουσία τη δημοκρατία, γιατί έτσι δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να σας ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σας έκθεση για το μέλλον της ΚΑΠ. Και ε, ταυτίζομαι με αρκετά σημεία της έκθεσής σας. Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει ουσιαστικά σε αυτά που ακούσαμε κατά τις προτάσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, γιατί Είπαμε από την αρχή ότι λείπει το όραμα, λείπει φιλοδοξία από τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ και φιλοδοξία ως προς τα γεωργικά εισοδήματα και ως προς τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιό μας, που αφορούν ε, την διατροφή, την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και το κλίμα. Και κατά τη γνώμη μου, η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά μια διοικητική μεταρρύθμιση ε, που υποτίθεται ότι ακολουθεί τις γραμμές της απλούστευσης και της επικουρικότητας, αλλά δεν είναι ουσιαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ενώ εμείς περιμέναμε για την περίοδο 2021-2027 μια πραγματικά ε, σημαντική μεταρρύθμιση για ένα μοντέλο μετάβασης της γεωργίας. Ε, αυτό όλα δείχνουν μια μεγαλύτερη δυσλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαίνεται και στο διαγωνισμό, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στο πι. Εκεί φαίνεται ε, μια ε, πολύ χαμηλή φιλοδοξία, πολύ χαμηλό επίπεδο φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΑΠΑ. Εσείς μιλήσατε για το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά αυτό το έχουμε ξαναδεί. Και με τη γαλακτοκομική κρίση, σα είχαμε πει κύριε Επίτροπε, έχουμε κρίση στο γάλα, θα πρέπει να παρεύετε. Εσεί μα είχατε πει, όχι, δεν, έχει, δεν έχουμε καμία κρίση. Και τώρα μου λέτε υπάρχει κρίση στο γάλα. Χρειάστηκε όμως ε, ε, να εξελιχθεί η κρίση και να έχουμε τεράστιες ζημίες μέχρι ότου αποφασίστε να επέμβετε και να τη ρυθμίσετε. Και παρόμοια κατάσταση έχουμε και τώρα. Φαίνεται, όπως λέει και η έκθεση, ότι αυτό το απλό γεγονός της επανεθνικοποίησης, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι μια φιλόδοξη απάντηση για την κοινή μας γεωργία. γιατί πρόκειται για στρατηγικές επιλογές που αφορούν την επιστηστική ασφάλεια ε, και η επιστηστική ασφάλεια σχετίζεται με την επιστηστική κυριαρχία. Φαίνεται ότι αυτό το ξεχνάμε με την επαρεθνικοποίηση. Και σίγουρα η πρόταση για τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων. Κύριε Φιγκερέντο, για το οικονομικό σκέλος, λέτε ότι οι άμεσε ενισχύσει δεν θα εγγυηθούν επαρκές γεωργικό εισόδημα. Και πιστεύω ότι το να συνδέσουμε το γεωργικό εισόδημα με την αποσύνδεση ή με τη στραματική ενίσχυση είναι λάθος. Γιατί θα μειωθεί ο γεωργικός προπολογισμό, οπότε θα μειωθούν και τα γεωργικά εισοδήματα. Θα πρέπει να είναι έρμη αυτής της πολιτικής η ε, γεωργή. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις αγορές και την κοινή οργάνωση αγοράς, ελάχιστα σημεία στην έκθεση αφορούν την ΚΟΑ και την κατάσταση στις αγορές. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, πληροφορίες. Επίσης, ποια είναι η σχέση της κοινή οργάνωσης αγοράς με τα στρατηγικά σχέδια. Γιατί έχουμε κάποια, α, κάποιους μηχανισμούς διαχείρισης των κρίσεων και ρυθμίσης αγοράς αλλά δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για τη διασύνδεση ΚΟΑ και στρατηγικών σχεδίων. Επίσης, τι γίνεται με την αγροτική πολιτική, την πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου. Γι' αυτό το σκέλος ε, ε, του γεωργικού προϋπολογισμού προβλέπονται δραστικές περικοπές. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι η αγροτική ανάπτυξη θα είναι το θύμα αυτών των περικοπών στο γεωργικό προϋπολογισμό. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Φιγκεραίδο. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Αν αξιολογήσουμε λίγο ουδέτερα την κατάσταση, είναι απόλυτα σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είχε κάποια καθήκοντα, τα ανέλαβε και ο Επίτροπος βεβαίως πρέπει μετά να απαντήσει. Για μένα ήταν κάπως ενοχλητικό το ότι μιλήσατε μόνο για ε, τις πληρωμές για τους τελικούς δικαιούχους από την πλευρά του συνεδρίου. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να μιλήσουμε ενσυνείδητα για οικογένειες γεωργών εδώ που παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα και όχι μόνο τρόφιμα, παράγουν και πολιτιστικές, έχουν και πολιτιστική απόδοση, οικονομική απόδοση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι μια πολιτική αξιολόγηση, μια ισορροπία πρέπει να βρεθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα και αυτό το delivery model της Κομισιόν στην ε, συζήτηση τελικά να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε. Έχω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί νομίζω, ε, επειδή δουλεύω με τον οριζόντιο κανονισμό, ότι υπάρχουν κάποια σημεία που χρήζουν διευκρίνησης σε σχέση με την ασφάλεια για την ε, ε, ε, για την απόκτηση γης. Μιλούσατε για, τις, για τους μηχανισμούς ελέγχου την, της Κομισιόν, για το κατά πόσο είναι επαρκής ή όχι. Ο ρόλος των αρχών πιστοποίησης ποιος είναι. Η πρόταση μιλά για τεράστια αύξηση των καθηκόντων προβλέπονται οι, μάλλον, οι διαδικασίες προβλέπονται αρκούν για να εξασφαλίσουν ότι οι απαραίτητες τεχνικές γνώσεις υπάρχουν. Και μιλάμε και για αυτά τα σχέδια δράσης, τα στρατηγικά σχέδια και όταν τα κράτη-μέλη ορίζουν μέσα σε αυτά τα ε, σχέδια, στόχους που ξεπερνούν το 25% πρέπει να εκπονήσουν και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Πόσο επαρκές και κατάλληλο θεωρείτε αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Γίνεται και κάποια αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτού για την επίτευξη των στόχων. Και επίσης μια εκτίμηση δική σας για για το ποσοστό ελέγχου και για τους, δύο, για τους δύο πυλώνες είναι διαφορετικό. Για τις άμεσες πληρωμές έχουμε 1% στον πρώτο πληρώνα, στην 5% ε, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτά τώρα θα συμπτυχθούν στις στρατηγικά, στα στρατηγικά σχέδια. Θα συμπτυχθούν και τα επίπεδα των ελέγχων. Και αν ναι, σε ποιο επίπεδο θα γίνει αυτό. Είναι τεχνικά τα ερωτήματα, αλλά τουλάχιστον για τη δική μου την έκθεση και για μένα είναι σημεία σημαντικά. Και επίσης η πολιτική αξιολόγηση που πρέπει να γίνει για το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε για τους γεωργούς. Αυτό είναι το δικό μας το καθήκον και αν ε, παραμείνουμε σε στενή συνεργασία και επαφή νομίζω ότι κάτι θα καταφέρουμε τελικά. Εγώ δεν είμαι τόσο επικριτική όσο άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα λοιπόν να ε, μου απαντήσετε σε αυτά. Ευχαριστώ. Μάλιστα, περνάμε στους συντονιστές τώρα. Ο κύριος από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φιγκερέιντο, που είστε σήμερα εδώ και μας παρουσιάζετε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ακούσαμε τα όσα μας είπατε για τη Γεωργία, για την χρηματοδότηση. Ε, έχουμε λίγο αντίθετες απόψεις βέβαια. Καλό θα ήταν να περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας γιατί είναι 40% το όριο για τους ε, γεωργούς στις, ε, ε, στην, για τη γεωργία. Πολλοί νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τελείως διαφορετικούς υπολογισμούς από τις Βρυξέλλες. Ίσως και αυτό να είναι μέσα στα καθήκοντά σας. Έχουμε δημόσιες δαπάνες 1% για 10 εκατομμύρια γεωργούς που φροντίζουν τα 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που έχουν. Ε, και μιλούμε για την παροχή τροφίμων σε μισό δισεκατομμύριο ε, ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει τα αριθμητικά στοιχεία λίγο να τα ξαναδούμε. Είναι σωστό αυτό για τους ε, γεωργούς. Μάλλον πρέπει να μιλήσετε και εσείς λίγο πιο ξεκάθαρα στο, στην κοινή γνώμη. Και έχω εδώ την άδεια οδήγησής μου. Το 61 στα 14 έβγαλα την άδεια οδήγησης. Τότε ε, την, ε, μου κόστησε κάποια 50 ευρώ, ας πούμε, με σημερινές τιμές. Αν δείτε την τιμή των σιτηρών του 61, τότε θα είχαν ε, δοθεί με τις σημερινές τιμές 30 δις παραπάνω για τους Γιώργους... θα είχαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ διαφορετικά ε, αριθμητικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς να, να δείτε τι γίνεται και με τις ε, ε μελέτες που υπάρχουν από την Βαβαρία εκείνης της εποχής για το πόσο έχουν προσφέρει η Βαβαροί ε, για το, και το πόσο τους έχει κοστίσει αυτό. Οπότε σας παρακαλώ σταματήστε να κατηγορείτε συνεχώς τους ε, γεωργούς. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την κοινή ε, γεωργική πολιτική. Θα το κάνουμε εμείς από κοινού και με την Κομισιόν. Ε, ξέρω τα συζήτηση που γίνεται για την εθνική ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε καλύτερα από τις Βρυξέλλες, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή λύση. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριο Καπούτο. Γεια σας κύριε Φιγερέτο. Ευχαριστούμε. Και καλώ ήρθατε και εσείς ε, κύριε ε, Χόγκαν. Ακούσαμε τώρα τι διαφορετικέ απόψεις για ε, το θέμα μας και τους δύο σας συζητούμε. Και εμείς ως συνομοθέτες όπως είπατε είμαστε στη μέση για να δούμε πώς θα βρεθεί η καλύτερη λύση. Ε, βεβαίως το ελεγκτικό συνέδριο κάνει τη δουλειά του, δηλαδή το να ελέγξει το να αξιολογήσει το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να σκεφτούμε ε, τις ε, ιδιομορφίες της ε, Εγώ θα εξέταζα λίγο περισσότερο την αποτελεσματικότητα των αμέσων πληρωμών και όλες τις δράσεις που αφορούν το περιβάλλον. Και οι δύο μας βεβαιώσετε για το πόσο σημαντική, πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας και ότι θα πρέπει και οι ε, πληρωμές να λάβουν υπόψη αυτές τις ιδιομορφίες. Οπότε θα πρέπει τα μέτρα για το περιβάλλον να συνδυαστούν με αυτή την ενισχυμένη αιρεσιμότητα. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την ε, κατεύθυνση που υποδεικνύεται. Και με τους ελέγχους που μας εξηγήσατε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Υπάρχει επίσης κανονικότης και ό,τι γίνεται να είναι νομότυπο. Σαν αμέσως επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε την μέση εδώ και γι' αυτό και σας ευχαριστούμε για όλα τα στοιχεία που μας εκθέσατε. Χόσλιν. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας, κύριε Φιγκερέιδο, γιατί πραγματικά μιλήσατε για την ουσία του πράγματος. Ο μεγάλος στόχος αυτής της μεταρρύθμισης λείπει και δεν προχωρούμε μόνο με τίτλους. Οι τίτλοι ωραία ακούγονται, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους ε, για το κλίμα κτλ. πρέπει να θέσουμε πολύ σοβαρά ερωτήματα. Οι Υπουργοί Γεωργίας ίσως καλά να το βρίσκουν αυτό, ε, γιατί ουσιαστικά καταργούμε την κοινή αγροτική πολιτική και αφήνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι νομίζουν. Η ελληνική έλεγχη επίσης είναι ένα προβληματικό σημείο. Αν η Γενική Διεύθυνση Άγκρη χάνει του μισού τη υπαλλήλου, δεν μπορώ να καταλάβω πώ θα γίνουν οι έλεγχοι βέβαια στα κράτη-μέλη, αλλά δεν γίνεται να αλλάζουν μόνο οι τίτλοι και τίποτε άλλο. Θα πρέπει πιο προσεκτικά να δούμε βεβαίω, γιατί αυτό που λέτε είναι ότι με τι άμεσε πληρωμέ θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια τροφίμων. Ε, λίγη σχέση έχουν άμεσε πληρωμέ ένα εκτάριο με την πιστιστική ασφάλεια, ωστόσο. Και μετά αν έχουμε πληρωμέ ανά εκτάριο, τι σημαίνει αυτό. Οι μισέ πληρωμέ, το λένε διάφορε μελέτε, ουσιαστικά πάνε στους, ε, ε, σε αυτούς που ουσιαστικά δίνουν την υγεία στους ε, γεωργού, που την ενοικιάζουν ή που την διαχειρίζονται. Οπότε τώρα με το 70% που έχουμε από τον πρώτο πυλώνα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Δεν ξέρω, μπορεί να, χρειάζεται, να χρειάζονται πήγοντα μέτρα για να δώσουμε περισσότερα κονδύλια στους γεωργούς. Και επίση αυτό που λέτε για τους στόχους για το κλίμα, που δεν, είναι, δεν μπορούν να επιτευχθούν με, την, με, το, με τον πρώτο πυλώνα. Πουθενά δεν το είδα εγώ αυτό γραμμένο. Βέβαια, εντάξει, καλό θα ήταν να με ακούγατε κιόλα όσο μιλάω. Δεν τελείωσα, πρόεδρε. Δεν τελείωσα, πρόεδρε. Ναι. Ήθελα να με ακούει ο κύριος Φιγερέιδο, γιατί είναι σημαντικό νομίζω. Πρέπει λοιπόν, όταν, όταν έχετε μια απέτηση για, τα, για το κλίμα, για το περιβάλλον, θα πρέπει να την περιγράφετε. Εδώ δεν περιγράφετε τίποτα. Είναι τόσο γενικόλογα όλα όσα λέτε που λέτε, εντάξει, αφ, αφ, γεωργοί κανονίστε τι θα κάνετε για το κλίμα και το περιβάλλον. Ε, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να μιλούμε για συγκεκριμένα πράγματα. Βιοπικιλότητα, κλίμα, περιβάλλον. Πρέπει πολύ συγκεκριμένα να μιλάμε για να είναι κατανοητά αυτά που ζητούμε δεν μπορούμε να λέμε οι μισές επιφάνειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βρίσκονται κάτω από αυτό το ε, περιβαλλοντικό μέτρο. Ούτε πρόκειται στο μέλλον αυτό να βελτιωθεί. Νομίζω ότι πρέπει να με ακούσετε προσεκτικά τι λέμε, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται αλλαγή η πολιτική σας. Ευχαριστώ. Θέλω να παραβαίνετε το χρονοβόλευσή σα. Περνάμε στι μονόλεπτε παρεμβάσει. Ο κύριο Κάρθη έχει το λόγο. Thank you, um, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πάρα πολύ θετικά μερικά στοιχεία από αυτά που ακούσαμε την έκθεση, ιδίω ε, ε, κάποιε διευκρινήσει όσον αφορά κάποια αριθμητικά στοιχεία. Τι γίνεται με τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Έχουμε περικοπή 15% γιατί αυτό το είχαμε ζητήσει και είπε όχι η Κομισιόν. Είναι η προβληματική του ΠΔΠ. Θα θελήσουν να βάλουν περισσότερα λεφτά τα κράτη-μέλη. Ενδιαφέρει πολλές χώρες. Πρόκειται για περικοπή πολύ σημαντική. Μπορεί να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο είδου άνω όριο όσον αφορά τις ε, πληρωμές και θα συνεχιστούν οι πληρωμές και δεν θα υπάρχουν τα παραθυράκια. Τώρα όσον αφορά τις ε, άμεσες πληρωμές είναι πολιτικό το θέμα και διαφωνώ με το Ελληνικό συνέδριο γιατί θέλουν να καταργήσουν αυτές τις άμεσες πληρωμές γιατί έτσι θα βγάλετε από τη μέση πολλούς γεωργούς και αυτό θα έχει επιπτώσεις για τα είδη διατροφής, την ποιότητά τους θα καταστραφούν πάρα πολλές κοινότητες, άρα θα πρέπει να τα ξανασκεφτείτε, να τα ξαναζυγίσετε τα πράγματα για τις άμεσες πληρωμές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω καμιά φορά πρέπει να μιλούμε και με εξωτερικούς θεσμικού παράγοντε ε, θεσμικούς παράγοντες, όπως το ελεκτικό συνέδριο. Ε, είναι σαφές ότι με τον πρώτο πυλόν έχουμε πρόβλημα. Η πρόταση του Επιτρόπου Χόγκαν προσπαθεί σε κάποια σημεία αυτό το πρόβλημα να το λύσει. Αλλά πολλά εκρεμή σημεία παραμένουν. Δύο ας πούμε. Αν τα κράτη-μέλη δεν σταματήσουν να χρησιμοποιούν το ιστορικό μοντέλο, θα πούν δύο ε, εκτάρια θα, πάρει, θα, θα πάρουν την τάδε ε, ενίσχυση ε, γιατί πριν από τόσα χρόνια είχε φυτέψει την τάδε καλλιέργεια. Δεν γίνεται να συνεχιστεί το σύστημα αυτό. Αν δεν το αλλάξουμε με σωστά κίνητρα και αν δεν βρούμε και μεταβατικές λύσεις, τότε δεν θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Στη δική μου την περιφέρεια υπάρχουν 3.000 εκτάρια από δέντρα όπου άνθρωποι που έχουν ε, α, απέτηση ε, για την, για την πληρωμή δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Με την προστασία του περιβάλλοντος τι γίνεται, με την, με την συμβολή για την προστασία του περιβάλλοντος. Μηδέν. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι σημαντικά προβλήματα του πρώτου πυλώνα. Αν αρχίζουμε, αν δεν δώσουμε χρήματα σε αυτούς που θέλουν και με καινοτόμο τρόπο να διαχειριστούν τις γέες τους από εδώ και μπρος, τότε θα έχουμε πρόβλημα, γιατί την, ε, κριτική του Ευρωπαίου φορολογουμένου θα την, έχουμε, θα την αξίζουμε. Ο κύριος Άγνιου. Είναι συναρπαστική αυτή η συζήτηση. Ε, η, πιο συζή... η ενδιαφέρουσα συζήτηση νομίζω που έχουμε κάνει ποτέ. Το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο, θεσμικό, ο μόνος ε, το μόνο θεσμικό όργανο που ε, σέβομαι. Γιατί μιλάμε πραγματικά γεγονότα στην Κομισιόν. 40% της ΚΑΠ του προπολογισμού θα πάει σε δράσεις για το κλίμα. Σημαίνει 20 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα προφανώ, όταν μιλάμε για τέτοιε δαπάνε, προφανώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά όταν ρωτάμε τι κάνει ο Γεωργό, είναι πολύ εύκολο ο Γεωργό να δείξει ότι κάνει αυτό που πρέπει θα πει ότι εγώ έχω σταματήσει να έχω 20% από την ε, αρωτρέα μου γη, δεν ε, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τα, τις παλιές καλλιέργειες, ε, κάνω εξοικονόμηση του διοξιδίου του άνθρακα, άρα έχω μικρότερα λίματα από την, από την καλλιέργειά μου, από την εκμετάλλευσή μου κτλ. Άρα εγώ έχω... βγάλει το τριφύλι από, τις, από τα χωράφια μου, οπότε δεν έχω μονοξίδιο του αζότου, όλα καλά. Πού πάμε όμως με αυτή την ε, νοοτροπία. Ο στόχος ήταν να βελτιωθεί το κλίμα. Αν θέλετε να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Τώρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, αντιμικροβιακή αντίσταση. Ε, θα μπορούσαμε να, έχουμε, να θέλουμε βιοασφάλεια για τις εκμεταλλεύσεις. Θα μπορούσαμε να βάλουμε χρήματα στην ε, ε, έρευνα για ε, κτηνοτροφία που μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ή να είναι όντως ανθεκτική. Θα μπορούσαμε να δώσουμε καλύτερα κορδίλια για καλύτερο εξαρισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τους δύο καλεσμένους μας επίσης. Η ΚΑΠ μετά το 2020 θα είναι ε, η ολοκλήρωση της αποτυχίας κοινή γεωρικής πολιτικής. Ήδη έχουμε σημαντική περικοπή του προϋπολογισμού, περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, επιμένετε στην απαραίτητη επικουρικότητα και θέλετε να ξαναδώσετε πίσω στις χώρες κάποιες εξουσίες. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να ικανοποιεί κάποιο που είναι υπέρ τη εθνική κυριαρχία, αλλά δεν είναι μένω ικανοποιημένο, γιατί περνάμε από μια ε, λογική τη υποταγή στο 95 που λέει ότι τα, οι πληρωμές θα γίνονται στα κράτη-μέλη ανάλογα με τα αποτελέσματα. Οπότε ισχύει ο ίδιος εκβιασμός και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα και τους ελέγχους, αυτό που είναι ανησυχητικό, πολύ ανησυχητικό θα έλεγα, γιατί δεν θα διορθώσει καθόλου τη, τη στρεβλώση του ανταγωνισμού και το ξέρετε, γιατί τα κράτη-μέλη ε, είναι ανήμπορα να δράσουν απέναντι στους οικονομικούς κανόνες που επιβάλλεται. Οπότε πώς θα λύσετε το βασικό πρόβλημα των γεωργών ε, και κυρίως ε, οι τιμές που θα λαμβάνουν για τα προϊόντα τους θα τους ανταμείβουν πραγματικά η ΚΑΠ μετά το 2020 θα σεβαστεί τους στόχου του άρθρου 39, στο οποίο αναφέρει στη συνέχεια, ε, ενώ στην ουσία δεν θα μπορέσετε να το εφαρμόσετε, την κατοχήρωση δηλαδή του γεωργικού εισοδήματος. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε το γύρο των συντονιστών. Περνάμε στου λοιπού ευρωβουλευτέ. Η κυρία Κατάινεν. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για την ε, διεξοδική μελέτη που μας παρουσίασε, παρόλο που διαφωνώ με τα βασικά πορίσματα της γνωμοδότησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ αξιόπιστη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε υπέρ μιας νέας προσέγγισης που θα δίνει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν ελεκτικά συστήματα και συστήματα παρακολούθησης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Δεν κρίνω απαραίτητο πέρα του νέου delivery model να έχουμε και ένα σύστημα αυστηρών ελέγχων βάσει του παλιού μοντέλου που υποτίθεται θα έπρεπε να είχαμε καταργήσει με τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντίθετα, θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να μειώσουμε τις διακητικές διατυπώσεις και σίγουρα δεν θέλουμε επικάλυψη με την εφαρμογή αυτού του διπλού συστήματος. Συμφωνώ ότι το σύστημα βάση επιδόσεων, βάση αποτελεσμάτων και οι δείκτες του θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω και οι βασικές ε, δράσεις θα πρέπει να αναλύονται πιο διεξοδικά. Επίση, ε, μόνο με μια αντίστοιχη επέκταση και σε άλλου τομεί. θα έχουμε μια αξιόπιστη λύση. Ευχαριστώ. κύριο Φλάνακαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Όλοι εδώ, ε, υποθέτω, θα ανατρίχεζαν στην ιδέα της περικοπής του γεωρικού προϋπολογισμού. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, οπότε δεν θα σας εκκλείσει η ιδέα ότι κάποιοι θέλουν να περικόψουν το γεωρικό προϋπολογισμό. Και θα έλεγα στα μέλη της Επιτροπής ότι ε, δεν συμφωνώ με όλη την έκθεση, αλλά κάποια στοιχεία λογικής ε, τα περιλαμβάνει. Και νομίζω λάθος θα ήταν να αγνοούμε τις προειδοποίησει, κυρίως τις προειδοποιήσει ότι μπορούμε σήμερα να πληρώνουμε γεωργούς για κάτι που είχαν κάνει πριν από 25 χρόνια. Και σίγουρα η τωρινή δομή σε αυτό το αποτέλεσμα θα οδηγήσει να ανταμείβονται άνθρωποι για κάτι που είχαν κάνει πριν από 25 χρόνια και να συνεχίζουν να λαμβάνουν ενισχύσει. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού κατηγορείται αυτή η η λογική και γι' αυτό προτείνεται περικοπή του προϋπολογισμού. Προσοχή λοιπόν. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται στην Επιτροπή Γεωργία. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα και αν κοφεύσουμε στι εκκλήσει των άλλων, θα μείνουμε με άδεια χέρια τελικά. Ευχαριστώ κύριε Ριμπέιρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φιγκερέντο, μας είπατε πολύ εύγλωτα ότι η ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, σε γεγονότα και όχι σε πολιτικές κρίσεις. Και ναι, μεν μας ε, δώσατε κάποια κριτήρια ελέγχου, απ' την άλλη κάνετε μια ανάλυση που μοιάζει αρκετά πολιτικοποιημένη. Γιατί αφισβητήσατε το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων και την ε, ύπαρξη του μακροπρόθεσμου οράματος της ΚΑΠ. Επίσης δεν προτείνεται καμία αλλαγή ούτε στο πεδίο εφαρμογή, ούτε στους στόχους ε, της ΚΑΠ. Οπότε τι προτείνεται να αλλάξει στο σύστημα άμεσων ενισχύσεων. Ε, δεν χρειάζεται μόνο γενική ανάλυση, θέλουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, όντως ίσως ε, υπάρξει πρόβλημα ελέγχου εξακρίβωσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Πού όμως έγινε το πρόβλημα που επισημαίνεται. Σε ό,τι αφορά τις ελεκτρικέ αρχέ, υπάρχει πρόβλημα ή το πρόβλημα οφείλεται στην περιπλοκότητα του συστήματος που επισημαινετε σε οτι αφορα τους εθνικες ελεκτικες αρχες υπαρχει προβλημα η το προβλημα οφειλεται στην περιπλοκοτητα του συστηματος που ειναι πολυ επιπεδο και δημιουργεί προβλήματα στα κράτη-μέλη. Και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του καινούριου και του παλιού μοντέλου που έχει παρόμοια στοιχεία ως προς το δεύτερο πλέον. Ευχαριστώ. Κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ απορρίπτω τη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου, την οποία κρίνω ιδιαίτερος πολιτικοποιημένη. Κανονικά θα έπρεπε να κάνετε κάποιες ε, αμερόληπτες ε, αναλύσεις και παρόλα αυτά εσείς προβαίνετε σε πολιτικές κρίσεις. Αμφισβητείτε ε, την το περιεχόμενο κάποιων πολιτικών. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε κατά πόσο τα κονδύλια δαπανώνται με βάση τους θεσμοθετημένους κανόνες ή αν έγινε κάποια κατάχρηση των κονδυλίων. Αυτό πρέπει να κάνετε τώρα για τις άμεσες ενισχύσεις. Τα βλέπετε όλα πολύ μαύρα άσπρα. Και δεν το λέω μόνο για τις άμεσες ενισχύσεις, γιατί οι άμεσες ενισχύσεις όχι μόνο είναι αποτελεσματικές και αυξάνουν το γεωργικό εισόδημα, αλλά αποτρέπουν και την απερίμωση των αγροτικών περιοχών. Οπότε θα πρέπει να δούμε τις, γενικές, τις ε, άμεσες ενισχύσεις στο γενικότερο πλαίσιο της γεωργίας και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, ε, λέτε έλεγχο γίνεται μόνο για τη μεταφορά κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη και όχι ε, εντό του κράτου-μέλου. Θα πρέπει να πλουστευτούν οι έλεγχοι και να γίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε Χόγκαν, όταν ε, ένα κάποιο επικριτικό σχόλιο του ανεξάρτητου φορέα του ελεκτικού συνεδρίου το απορρίπτεται έτσι ε, νομίζω ότι το ε, ελεκτικό συνέδριο έκανε την δουλειά του με βάση συγκεκριμένα ε, δεδομένα. Θα πρέπει ίσως να δείτε λίγο πιο προσεκτικά τα όσα λέει. Κύριε Φιγκερέιντο, μπορείτε κάπου ίσως να δείτε πού υπάρχουν αυτές οι παρανοήσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού έχει γίνει η παρεξήγηση. Και επίσης για την επανεθνικοποίηση, ε, το ότι θα έχουμε πρόβλημα για τα διάφορα κράτη-μέλη που θα έχουν διαφορετικά πρότυπα και θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική αξιολόγηση, είναι δύσκολο να δούμε πώ θα μπορέσουν να τηρηθούν οι στόχοι. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία πολύ καιρό την κάνουμε. σω θα μπορούσατε να τη σχολιάσετε. Και επίσης ε, σε σχέση που, με αυτό που είπε και ο συνάδελφος Ντες, ε, είναι πριν από την ε, ε, ΚΟΑ, ωστόσο, η, περίοδος που περιγράφεται. από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ευχαριστώ κύριο Σταραμπέλα. Ευχαριστώ. Κύριε Φιγκερέντο, κύριε Επίτροπε. Και εγώ εκτιμώ την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που επισημαίνει κάποιες αντιφάσεις και τον τρόπο που εφαρμόζουμε τις ενισχύσεις που δεν κατανέμονται σωστά ανάλογα με τις ανάγκες των ε, γεωργών. Γιατί άλλοι λαμβάνουν ε, δαψιλές ενισχύσεις και άλλοι πολύ φιδωλές. Ε, και έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ορισμένοι γεωργοί. Επίσης, αμφισβητείτε τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων που είναι στρεματικές. Συμφωνώ με την επικριτική που ασκείται. Εγώ ενδιαφέρομαι για το δεύτερο πυλώνα. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις πέραν της δικής σας που να δείχνουν ότι υπάρχουν κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται, υποχρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται εσφαλμένα. Γιατί σε πολλές χώρες δεν φτάνουν τα κονδύλια στις αγροτικές ζώνες. Γιατί ε, γίνεται υπεξαίρεση τους, χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς ή δεν χρησιμοποιούνται επειδή δεν υπάρχει το απαραίτητο ποσοστό σε χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για τις ομιλίες τους. Έχουμε επιμείνει στο θέμα των ελέγχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γιατί διαπιστώσαμε πόσο παράλογο είναι το σύστημα όταν ε, ασκεί έναν υπερβολικά λογιστικό έλεγχο των στρεματικών ενισχύσεων και ε, μερικές φορές ε, ε, δύο τετραγωνικά μέτρα ακριβώ επειδή τα έχουν πατήσει αγελάδες μπροστά στο μέρος που ποτίζονται θεωρούνται ότι δεν αξίζει να, να συμπεριληφθούν στη στρεματική ενίσχυση. Επίσης, εμείς ε, έχουμε το νέο delivery model που κλείνει με βάση τα αποτελέσματα και όχι με βάση τους περιορισμούς. Αντιλαμβάνουμε τις επιφυλάξεις για την πολιτική που στηρίζεται μόνο στα αποτελέσματα, αλλά για ποιους λόγους ε, ότι θα πρέπει να προσέχουμε σε αυτή τη μετάβαση προς μια πολιτική των αποτελεσμάτων και όχι των μέσων. Επίσης λέτε ότι με τη μορφή που έχει πρόταση δεν ε, επιτρέπεται η πιστοποίηση της κανονικότητας και της νομιμότητας του συνόλου των δαπανών. Τι αλλαγέ λοιπόν προτείνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην πρότασή της για να καλυφθούν οι ανησυχίες σας, η κυρία Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ και του δύο για τη συζητήσει σα παρατήρηση. Θα ήθελα πάρα πολύ το ηλεκτρικό συνέδριο να δει τους σκοπούς της ΚΑΠ και να δει το πρόβλημα του εισοδήματος των γεωργών, το πρόβλημα του περιβάλλοντος και αυτά να τα αποτιμήσει οικονομικά και έτσι να έχουμε έναν προπολογισμό που να βοηθάει στο έργο μας. Αν τα παρουσιάζετε και τα αναλύετε έτσι, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένη. Πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης τελικά τι γίνεται μακροπρόθεσμα, ποιο είναι το όραμά μας, γιατί τελικά ε, η πραγματικότητα του προπολισμού μας ε, φρέναρει επίσης όσον αφορά το δεν έχουμε κάποια στεγανά στοιχεία για τον ρόλο των ε, αμέσων πληρωμών. Δεν πήγαινε να ρωτήσετε τους γεωργού στην εκλογική περιφέρεια που για το εισόδημά τους σε αυτέ τις πληρωμέ στηριζόνται και τώρα απειλούνται από τις περικοπές. Για κοιτάξτε τους στόχους της ΚΑΠ και το ότι οι γεωργοί θέλουν να πετύχουν το στόχο που αφορά το περιβάλλον. Θέλουν, αλλά δεν βοηθάει ο τρόπος που τσακώνεστε με τη Γενική Διεύθυνση της ε, Κομισιόν. Μην τα συζητάμε εκ των υστέρων, δεν χρειάζονται κουβέντες, χρειάζεται προσανατολισμός. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το ελληνικό συνέδριο. Και εγώ Θέλω να χαιρετήσω την εκθεσή σας, γιατί μας υποστηρίζει στη δική μας δουλειά. Ε, διαφωνώ με τον κύριο Ντε. το θέμα δεν είναι ε, τι θα κάνουμε με την, με την ε, Γεωργία. Το θέμα είναι πώς θα δώσουμε τα κονδύλια, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτερα τι γίνεται στους γεωργού. Ακριβώς για τους γεωργού είναι σημαντικό γιατί θέλουμε να είναι ανθεκτικές οι ε, εκμεταλλεύσεις και για τα όσα αφορούν στο περιβάλλον, για την εκτινοτροφία, για τις κοινέ γεωργικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν με σωστό και στοχευμένο τρόπο για να βοηθήσουμε τους γεωργούς και αν δούμε τώρα τις τιμές του 1961, αν θέλουμε να έχουμε αυτές τις τιμές, ε, πρέπει, να έχουμε, πρέπει να καταργήσουμε την υπερπαραγωγή και τις εξαγωγές. Ο κύριος Κολομπία. Ευχαριστώ. Επ' ευκαιρία της συζήτησης ε, επί της του ελεκτικού συνεδρίου ε, ρωτάμε κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν σωστά τα κονδύλια. Για τι άμεσε ενισχύσει, χάρη σε αυτές θεωρητικά ζουν αξιοπρεπώς οι Γεωργοί, θεωρητικά και το τονίζω, αλλά η πραγματικότητα αλλιώ έχει. Ε, πριν από μερικές εβδομάδες πήγαμε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Βουλγαρία Εκεί για τρεις ώρες συναντηθήκαμε με εθνικούς ηθήνοντες ε, από το γεωργικό κλάδο και με προσώπους του Υπουργείου Γεωργίας. Μας είπαν κάτι που ήταν ανατριχιαστικό και αυτή είναι η πραγματικότητα. 80% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνουν στο 6% των γεωργών στη Βουλγαρία. Και Υφυπουργό τη Γεωργία μα μίλησε για 85% των ενισχύσεων που ωφελούν 10% των γεωκτημόνων και όχι ε, τους γεωργούς, όχι αυτούς δηλαδή που καλλιεργούν τη γη, αλλά στους γεωκτήμονες πηγαίνουν ε, οι άμεσες ενισχύσεις. Και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Και μάλιστα στην Βουλγαρία έχουμε 350.000 οικογενειακές εκμεταλλεύσεις κάτω των 5 εκταρίων. Και εκεί ο αντίκτυπο των άμεσων ενισχύσεων ποιο θα είναι, γιατί με τη μείωση του γεωργικού προπολογισμού θα μειωθούν ακόμη περισσότερο τα εισοδήματα τους. Α το σκεφτούμε λοιπόν και θα αλλάξουμε μέθοδο. Νόιχλ. Ευχαριστώ. Στο γραφείο σας παρακολουθούσα και είχα, έχω ένα μια ερώτηση προς το ε, εκλεκτικό συνέδριο. Καταρχάς ευχαριστώ για την έκθεση. Για άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπάρχουν ε, τέτοιες πληρωμές σε αυτό το ύψος. Υπάρχουν άλλοι τομείς, οικονομικοί τομείς της Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχουν ε, τέτοιες ε, πληρωμές συνδεδεμένες με τις, με τις με τις επιφάνειες. Και αν υπάρχουν τέτοιες κοινωνικές, ας πούμε, πληρωμές, οι, μπορούν να επιβιώσουν αν, υπάρχει, αν αυτό που δίνουμε στους γεωργούς είναι κοινωνική επιδότηση, υπάρχουν άλλα ευρωπαϊκά παραδείγματα κοινωνικών επιδοτήσεων που χωρίς να ελέγχονται γίνονται, καταβάλλονται χωρίς να είναι σαφές εάν κάποιος έχει ανάγκη για, αυτή την, για αυτό το επίδομα ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Είχαμε πολύ καιρό να παρακολουθήσουμε τόσο σφοδρή συζήτηση και τόσο ζωηρή και τόσο ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε λίγο, αλλά χαλάλη. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, πρώτα στον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Φιγκερέντο και μετά στον Επίτροπο Χόγκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμότατα για τις ερωτήσεις που διατυπώσατε. Και χαίρομαι που η γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου προκάλεσε τόσο ζωηρή, τόσο ζωντανή συζήτηση. αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερος. Φοβούμαι ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, γιατί ήταν τόσες, τόσο πολλές. Μερικές φορές βέβαια επαναλήθηκαν, από διάφορες πολιτικές ομάδες, αλλά ήταν παρόλα αυτά πολύ άριθμες. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας, μπορώ πολύ ευχαρίστως να έρθω και άλλη φορά στη συνεδρίασή σας για να απαντήσω πιο διεξοδικά στις ερωτήσεις σας. Τώρα έχω μόνο ένα δεκάλεπτο και αν μου επιτρέπει ο πρόεδρος θα μιλήσω πρώτα εγώ και μετά θα ζητήσω τον, από τον άλλο συνάδελφο του ελεκτικού συνεδρίου να απαντήσει στις πιο τεχνικές ερωτήσεις. Δέκα λεπτά συνολικά, λέει ο πρόεδρο. Καλώ, είμαι πολύ λακωνικό στι απαντήσει μου. Καταρχήν, ω προ τα γενικά σχόλια του αξιότιμου επιτρόπου, θα ήθελα να πω ότι είναι αλήθεια ότι από τον Ιανουάριο συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Ιανουάριο οι υπηρεσίε του Ελεκτικού Συνεδρίου και του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντιόνται και συζητούν. Και τον Ιούνιο ενημερωθήκαμε για τις προτάσεις. Και ήταν σαφές από τις συναντήσεις μας ότι είχαμε πολλές αμφιβολίες. Από την αρχή τις επισημάναμε ότι είχαμε πολλές αμφιβολίες για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε, η τελική μας γνωμοδότηση δεν θα πρέπει να ευνηδιάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί από την αρχή είχαμε επισημάνει τις αμφιβολίες μας. Και όταν έλαβα την επιστολή του Επιτρόπου Χόγκαν στις 16 Οκτωβρίου, τη διάβασα πολύ προσεκτικά και οφείλω να πω ότι τα επιχειρήματα που παρέθεσε την επιστολή του μας ήταν ήδη γνωστά. Γιατί είχαμε ήδη ξεκινήσει τη συζήτηση σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ Ελεκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ τη μορφή ότι παρεξήγησα τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, τις μελέτησα όσο πιο διεξοδικά γινόταν. Τις διάβασα κατά λεπτού και με τον και με το σίγμα δεν υπάρχει περίπτωση να τις παρεξήγησα. Και τα σχόλιά μου είναι χαρακτηριστικά της αναλυτικής μελέτης ε, της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες. Αυτό που λέμε είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τελικά. Γιατί οι εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τις επιλογές των κρατών μελών για τα περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, εξαρτώνται από την αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Εθνικών Επιλογών. Οπότε δεν ξέρουμε τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αξιολογήσεις των επιλογών των χωρών μελών. Κάτι άλλο που λέμε στη γνωμοδότηση είναι πώς μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η συμβολή των δαπανών της ΚΑΠ για τα περιβαλλοντικά θέματα θα είναι 40% όταν οι τρέχουσες περικοπές είναι 19,6% και είδαμε στους ελέγχους μας ότι ούτε αυτός ο έλεγχος δεν είχε, ούτε αυτός ο στόχος δεν είχε υλοποιηθεί, το 19,1%. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να τηρήσουμε το 19%, πώς να πιστέψω ότι θα τηρήσουμε το 40%, πώς θα δικαιολογηθεί αυτό το άλμα από το 19% στο 40% είμαι υποχρεωμένο ω να επισημάνω αυτή την αδυναμία κατά τη γνώμη υλοποίηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τι άμεσε ενισχύσει, θα πρέπει και εδώ να είμαι σαφή. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι υπέρ ούτε κατά των άμεσων ενισχύσεων. Δεν είναι αυτό το θέμα. Οι άμεση ενισχύσει είναι πολιτική επιλογή. Από τη στιγμή όμω, που οι συνομοθέτε λαμβάνουν την απόφαση να διατηρήσουν ως βασικό εργαλείο της ΚΑΠ, της άμεσες ενισχύσεις, που μάλιστα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% του προϋπολογισμού, τα οικονομικά στοιχεία αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι σαφή. Και για μένα είναι σαφές ότι τα οικονομικά θεμέλια αυτής της επιλογής δεν είναι σαφή. Γιατί ακόμη και εσείς είστε διχασμένοι μεταξύ σας. Δεν υπάρχουν οικονομικά πιστήρια που να συνηγορούν υπέρ της διατήρησης των άμεσων ενισχύσεων. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά των άμεσων ενισχύσεων. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτό που σας ζητώ είναι να μας παρουσιάσετε τις οικονομικές ενδείξεις, τα οικονομικά πιστήρια που να στοιχειοθετούν αυτή σας την επιλογή. Και κυρία Ράς Γκαρσία, εγώ δεν προτείνω κατάργηση, ούτε επιτίθεμαι μάλλον στις άμεσες ενισχύσεις. Κύριε Κάρθη, δεν επιτίθεμαι στις άμεσες ενισχύσεις. Ούτε είναι πολιτική μου η κρίση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πολιτικοποιημένη η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Και κάτι άλλο. Μία παρατήρηση που έγινε από τον Επίτροπο Χόγκαν. Είπε ο Επίτροπος ότι η δημοσιονομική διαχείριση στις αγροτικές ε, περιοχές ήταν πολύ επιτυχημένη. Όντως. Και το είπαμε κι εμείς. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο το είπε στην ετήσια έκθεση πριν από δύο εβδομάδες, πριν από τρεις εβδομάδες, είπαμε αυτό το στοιχείο, ότι όντως έχουμε βελτιώσει πολύ τη δημοσιονομική διαχείριση, προκειμένου να επιτύχουμε τα καλά αποτελέσματα. Και μάλιστα χρησιμοποίησαμε όλους τους μηχανισμούς που είχαμε στη διάθεσή μας. Και αυτό που λέει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο είναι ότι όταν κάνουμε μια κίνηση και όταν κάνουμε κάποια αλλαγή, δεν μπορούμε με την κίνηση και την αλλαγή αυτή να θέτουμε σε κίνδυνο τα προηγούμενα επιτέγματα. Εγώ δεν σας ζητώ να θεσπίσετε περισσότερους ελέγχους. Δεν σας ζητώ να αυξήσετε το διοικητικό φόρτο και να επιβάλλετε περισσότερες διοικητικές διατυπώσεις στους γεωργού. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γιατί οι κανονισμοί δεν παραδέχονται ότι όλες οι δαπάνες θα πρέπει να τηρούν το ενωσιακό δίκαιο. Γιατί μόνο το 2% των δαπανών απαιτείται να τηρεί το ενωσιακό δίκτυο και αυτό ελέγχεται. Και οι αρχές πιστοποίησης, όταν θα επιτελούν το έργο τους στα κράτη-μέλη και θα ελέγχουν την ομιμότητα και την κανονικότητα, θα το κάνουν μόνο και το 2% των δαπανών. Γιατί λοιπόν αυτές οι αρχές πιστοποίησης δεν θα μπορούν στο μέλλον να ελέγχουν το σύνολο των δαπανών και το υπόλοιπο 98% δηλαδή. Και δεν σας το ζητάει αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Εγώ σας ρώτησα, γιατί απαιτείται κάτι τέτοιο στο γενικό δημοσιονομικό κανονισμό και δεν το απαιτείται ταυτόχρονα από τις δαπάνε τις γεωργικές που είναι ένα μεγάλο ποσοστό του κοινοτικού προϋπολογισμού διαπιστώνω μια αντίφαση εδώ ω ελεκτή. και οφείλω να την επισημάνω κύριε Μπούντα οι ελεγκτές δεν παρακολουθούν μόνο που πάει το χρήμα αλλά το κάνουν την ώρα, τη στιγμή που κάνουν το λογιστικό έλεγχο άλλα δύο λεπτά λέει ο Πρόεδρος εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να επιστήσουμε την προσοχή του νομοθέτη στις συνέπειε που θα έχουν οι νομοθετικέ τους επιλογές. Δεν θα υπαγορεύσουμε εμείς κάποιε επιλογές, εμείς θα παρακολουθήσουμε την πορεία του χρήματο. Και φυσικά θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες που θα θεσπίσετε. Αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή που θα το κάνουμε. Θα δώσω το λόγο στον Πίτερ να κάνει κάποια τεχνικά σχόλια, που έχει δύο λεπτά. Η κυρία Ρώτησε τι γίνεται με τα σχέδια δράση που προβλέπονται. Αν θυμάμαι καλά, αυτά θα ξεκινήσουν εάν υπάρξει απόκληση μεταξύ του αποτελέσματο και του σχεδίου, πάνω από 25% που είναι σημαντική απόκληση. Ε, είναι σημαντική η ερώτησή σα, γιατί νομίζω ότι θα εξαρτηθεί ακριβώ η επιτυχία του project αυτού από, την, ε, ε, από το κατά πόσο θα υπάρξει ανάγκη για ένα σχέδιο δράση αλλά σίγουρα θα υπάρξει αρκετός χρόνος ε, για τα κράτη-μέλη για να απαντήσουν σε όλα αυτά. Ε, οπότε αναρωτιέμαι αν μπορούν να απαντήσουν μέσα στο ε, χρονικό όριο που έχουν. δεν ξέρω αν μας είχε ζητήσει κάποιος να μιλήσουμε για τον χαμηλό για το χαμηλό ποσοστό σφάλματος ευχαρίστως να το αναφέρουμε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ε, μίλησα για τον, για το ποστό λάθος, γιατί καμιά φορά θέλουμε και εμείς να ακούμε ένα κοπλιμέντο ε, σε σχέση με την ε, ΚΑΠ. Είμαστε στο 2,2%. Ε, νομίζω ότι το σύστημα που έχουμε δουλεύει καλά ακριβώ λόγω τη ε, δουλειά που κάνουν και οι συνομοθέτε και οι οργανισμοί πληρωμών των κρατών μελών. Οι άμεσε πληρωμέ είναι όντω πολιτικό μέτρο, όπω είπε ο κ. Φιγκεραίδο και στην ε, έκθεσή του, και δεν υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία ω προ αυτό. Η Κομισιόν λοιπόν δίνει αυτά τα στοιχεία, τα οποία αγνοήθηκαν πλήρω και παντελώ. Όσο περισσότερο βάλει κανεί στη βασική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερα μέτρα και παρεμβάσει χρειάζεσαι. Και μετά χρειάζεσαι ε, κριτήρια, αξιολόγηση, κριτήρια επιλεξιμότητα, κατευθυντήρε γραμμέ. Και μετά πρέπει να ελέγξει όλα αυτά που έχει θεσπίσει. Γι' αυτό δημιουργείται η γραφειοκρατία. Αυτό ακούω συνέχεια από τα κράτη-μέλη και από γεωργού. Πρέπει να καταργήσετε αυτή τη γραφειοκρατία. Και γι' αυτό κάνουμε μια απόπειρα με αυτή την ε, πρόταση να την καταργήσουμε. Αν τώρα ε, έχετε ε, αντιθέσεις, αντιρρήσεις, έχετε πολλές ευκαιρίες να μας τις αναφέρετε. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ την πρόταση της Κομισιόν, Πρόεδρε, απλώς θέλω να δούμε το πώς ε, παρουσιάστηκαν αδίκως ε, ή λαθασμένα αυτά που ανέφερα για την έκθεση του ε, Ελεκτικού συνεδρίου. Το Ελεκτικό συνεδρίο έχει τη δική του δουλειά, εγώ έχω τη δική μου δουλειά. Και βεβαίω και το κολέγιο των επιτρόπων μπορεί να σχολιάσει με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Δεν έχω ιδέα σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν υπόψη στο μέλλον από οποιαδήποτε έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου τα σχόλια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω εσεί θα δείτε την πρόταση Κομισιόν, θα δείτε και την έκθεση του συνεδρίου. Είχατε την ευκαιρία να κάνετε και την ε, ανταλλαγή απόψεων ε, ε, για την έκθεση του εισηγητή σα για την έκθεση τη Κομισιόν και μετά ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για το μέλλον. Και βεβαίω εμεί προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία μα τι επόμενε εβδομάδε, του επόμενου μήνε και αργότερα για να δούμε πού τελικώ θα καταλήξουμε. Αλλά οι γεωργοί μα χρειάζονται ασφάλεια, προβλεψιμότητα και πρέπει να τους το δώσουμε αυτό μέσω των ε, διαβεβαιώσεων που θα υπάρξουν από τους πολιτικούς. Ε, βεβαίως και το, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις σε πολλά θέματα και αυτό το αναμένουμε. Έτσι διεξάγεται η πολιτική διαδικασία. Αλλά να πω ότι το Μάρτιο του 2018 το Ελεκτικό Συνέδριο υπέβαλε μια έκθεση για το μέλλον της ΚΑΠ που ήταν ως απάντηση στην ανακοίνωση της Κομισιόν του Νοεμβρίου του 2017 και έτσι καθορίστηκαν οι βασικέ αρχέ για το τι περιλαμβάνει η νομοθετική πρόταση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Μετά από πολλέ συναντήσει με το ελεκτικό συνέδριο και ανταλλαγέ απόψεων, δημοσιεύθηκε αυτή η έκθεση. Και δεν θυμάμαι το ίδιο επίπεδο λεπτομερού κριτική που είδα σήμερα για την ε, έκθεση αυτή, από την έκθεση αυτή για την νομοθετική πρόταση. Οπότε εμεί δεν είχαμε καμία ιδέα ότι είχατε τόσε πολλέ ανησυχίε και προβλήματα για την τελική έκθεση. Δεν, είχα, δεν μας το είπε κανένας, δεν μας το ψιθύρισε κανένας αυτό. Ίσως εμείς δεν καταλάβαμε κάτι, αλλά δεν είχαμε πραγματικά κανένα δείγμα. Τέλος πάντων ούτε η υπηρεσία μου ούτε εγώ κατάλαβα να υπάρχουν ε, τόσες πολλές αντιρρήσεις τις τελευταίες δέκα φορές που συναντηθήκαμε. Τώρα για το νέο delivery model και για την νομιμότητα και την τακτικότητα των ε, πληρωμών. Αυτό, το, αυτό είναι ένα σύστημα που δίνει μια εναλλακτική λύση για το σύστημα που ήδη έχει, έχει κατακριθεί από πολλούς. Ότι είναι πολύ περίπλοκο, ότι δεν, ότι δεν επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και την απόδοση. Τώρα έχουμε μια πρόταση που θέλει να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα και την απόδοση και πάλι ακούμε επικριτικά σχόλια. Ο κύριος Άγνιου και ο κύριος Φιγκερέιδο και εμεί και είμαστε σε συμφωνία. Ο κύριο Άγγλου δεν συμφωνεί ούτε με τον κύριο Φιγκερέιδο ούτε με μένα. Αλλά οι προτάσει που υποβάλαμε καταστούν σαφέ ότι το νέο σύστημα θα βασίζεται στα αποτελέσματα και την απόδοση. Και όλοι οι δείκτε, όλοι οι στόχοι, όλε οι παρεμβάσει θα περιλαμβάνονται στη βασική πράξη. Αυτό λέει η νομοθετική πράξη. Η νομοθετική πρόταση, συγγνώμη. Ίσως να μην το έχετε διαβάσει επαρκώ. Αλλά όλα αυτά τα θέματα που αναφέρατε θα πρέπει να μπουν στην βασική ε, νομική πράξη και βρίσκονται στην πρόταση που ε, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο. Τώρα τι κάνουμε. Βλέπουμε ότι οι έλεγχοι από ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προσπαθούν, ε, καταστρέφονται ουσιαστικά. Ε, οπότε προσπαθούμε να έχουμε ένα σύστημα που να έχει όντω ε, καλού ελέγχου και να βασίζεται στην απόδοση και τα αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με του ε, κανόνε. Δεν, δεν θεωρώ ότι αν παρεκκλίνουμε βέβαια και λίγο από του κανόνε μπορεί να καταστραφεί ο κόσμο. Προσπαθούμε να, προσπα, να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια Και βεβαίω θέλουμε και τα κράτη-μέλη από τη δική του πλευρά να κάνουν τη δική του δουλειά. Θέλουμε να είναι πιο στοχευμένη η προσέγγιση μα και τα κράτη-μέλη να, να δουν ότι αυτές, αυτά που μας ζητούν τόσα χρόνια για να μπορούν να κάνουν περισσότερα για τους, για τους ε, ε, γεωργού του με λιγότερη περιπλοκότητα θα μπορούν να το κάνουν τώρα με αυτή την πρόταση. Οπότε ο ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό γίνεται σύμφωνα με τις κοινέ απαιτήσει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα και με την προσέγγιση για του νέου ελέγχου. Οι οργανισμοί πληρωμής θα είναι αυτοί που θα πρέπει να συμμορφωθούν με τι βασικέ απαιτήσει. Είχατε πει ότι οι ε, οργανισμοί πιστοποίηση δεν ήταν αξιόπιστοι. Θα υπάρξουν διορθώσει στι μεγάλε ελλείψει που υπάρχουν από τα συστήματα των κρατών μελών. Αυτό δεν διαφέρει από το τι γίνεται τώρα. Απλώ θα υπάρχουν λιγότεροι ευρωπαϊκοί κανόνε. Και θα υπάρχουν και θα βασίζονται στι μεμονωμένε συναλλαγέ. Αλλά το ε, ε, ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να λέει ότι υπάρχει ένα 2% με 98% σε αντίθεση με 98%. Ε, ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε να απαντήσω και ευχαριστώ κύριε Φιγκερέντο και κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για την ευκαιρία που είχαμε σήμερα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ε, Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αν και δύσκολη, αλλά σίγουρα απαραίτητη, γιατί τώρα ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής. Είναι από τα πιο περίπλοκα και δύσκολα ζητήματα πολιτικής γεωργία και εμπλέκονται και πολλά θεσμικά όργανα και πολλοί μηχανισμοί και φυσικά τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ε, μπορεί ε, να ασκήθηκαν κριτικές ακόμη και επικρίσεις από το ελεκτικό συνέδριο, αλλά ταυτόχρονα ακούσαμε και πολλές σκέψεις και προτάσεις ε, στη συζήτηση. Γι' αυτό και η δική μας Επιτροπή, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Άγκρη και ε, ο αρμόδιος επίτροπος θα τα εξετάσουν όλα αυτά πολύ ενδελεχώς. Ε, μερικές φορές είμαστε πολύ αυστηροί ε, απέναντι στην κοινή γεωργική πολιτική και περιμένουν πώς και πώς αυτές οι επικρίσεις οι πολέμοι της ΚΑΠ γιατί είναι νερό στο μήλο τους. Ε, ενώ εμείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη το συμφέρον των γεωργών μας και να είμαστε κριτικοί επί της ουσίας, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουμε και λίγο το μέτρο στην κριτική μας. Γιατί το μεσημέρι μου και σε μια άλλη συνάντηση που άκουσα ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ΚΑΠ και μερικοί περιμένουν πώς και πώς για να περιορίσουν την κοινή γεωρική πολιτική. Δεν θα πρέπει όμως η δική μας επιτροπή να συμβάλλει ενισχύοντας τα επιχείρηματά τους και να συμβάλλουμε στη μείωση της γεωρικής πολιτικής του γεωρικού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ τους καλεσμένους μας. Παρατείναμε αρκετά την ε, πρώτη μας συζήτηση λόγω του ενδιαφέροντος που είχε, αλλά έχουμε και άλλα θέματα. Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Φαντάζομαι όμως θα συνεχιστεί η συζήτηση μεταξύ μας και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ συνεργασία που έχουν τα θεσμικά μας όργανα. Ακόμη και μεταξύ φίλων ακούγονται ε, πολλές φορές επικρίσεις, αλλά μεταξύ φίλων επιτρέπονται ακόμη και τέτοια κριτικά σχόλια. Ευχαριστώ θερμά και τις ε, οι ε, συγκεκριτέ μας και τώρα ετοιμάζεται και ο τη επόμενη έκθεσης, ο κύριο Αντριέ. Θα πρέπει αμέσω να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το σημείο 8, που προβλέπει η συζήτηση της έκθεσης του κύριου Αντριέ. Σας θέρμα παρακαλώ να με βοηθήσετε γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρόνο. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τους χρόνους ομιλίας. Ο κύριος Αντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία παρατήρηση μου επιτρέπετε. Δεν νομίζω ότι ήταν χαμένος ο χρόνος που πέρασε. Δεν το χάσαμε το χρόνο μας τον αναλώσαμε σε πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και χάρη στην προηγούμενη συζήτηση θα διευκολύνω θα διευκολύνουμε και την παρουσίαση της δικής μου έκθεσης που βρίσκεται και αυτή στην καρδιά του προβλήματος. Πριν σας παρουσιάσω την έκθεσή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με βοήθησαν και φυσικά τους βοηθούς μου, το γραφείο μου, τον Αλεξάνδρ και τη Φραντσέσκα από τη Γραμματεία της Επιτροπής Γεωργίας και φυσικά και τη Μάγκη και των Μύρων, τους βοηθούς της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτό το συλλογικό έργο που κατέληξε στην έκθεση. Η έκθεσή μου παρτίζεται από τέσσερα τμήματα. Γιατί ξέρετε ότι τροποποιήθηκε το πλαίσιο της κοινή οργάνωσης αγοράς και το είδαμε και στην πρωινή συζήτηση ότι έγιναν κάποιες αλλαγές. Εγώ θα σας προτείνω το τμήμα της ενίας ΚΟΑ που αφορά κυρίως τον αμπελονικό τομέα ε, κατόπιν θα σας ε, αναφέρω τα ζητήματα ποιότητας που πραγματεύεται η έκθεση και τρίτο θέμα τα ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές και τα νησιά του Αιγαίου και τέταρτο τμήμα της έκθεσης προτάσεις της Επιτροπής που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησής μας γιατί προτείνουν παρέμβαση απέναντι στην απορρίθμιση και στην μεγάλη αστάθεια των τιμών. Σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα τη ενιαία ΚΟΑ, που αφορά κυρίω τα εμπελονικά ζητήματα. Πολύ σύντομα, μια και μου το ζητάτε, κύριε Πρόεδρε, για τον τομέα του ίνου. Ε, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έξι σημεία γρήγορα. Συμφωνώ με την ανάγκη να βελτιώσουμε την ελαστικότητα στη μέθοδο ε, υπολογισμού των ε, επιφανειών για την αδειοδότηση για τις νέες καλλιέργειες. Επίσης, ε, διαγράφουμε την προθεσμία του 2030 που προβλέπεται για να σταματήσουν για να σταματήσει το καθεστώς έγκρισης και να περάσουμε σε μια αποκεντρωμένη διαχείριση του καθεστώτος και αυτό το υποστηρίζω στην έκθεση. Δεύτερον, διεύρυνση των ποικιλιών και εκεί συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρήση ε, κάποιοι, της βήτης μπρούσκα και, ε, αφήν, και λαμβάνουμε υπόψη τις πέντε απαγορευμένες ε, ποικιλίε και έτσι ε, διευρύνουμε τη βιοπικιλότητα και προσαρμόζουμε το αμπέλι στις κλιματικές αλλαγές. Δεδομένου ότι αυτές οι επιλογές και αυτές οι χρήσεις θα εξαρτηθούν από την ε, βούληση των κρατών μελών αλλά και των ε, αμπελουργών, γιατί πρόκειται για ένα προαιρετικό πλαίσιο, ένα θελοντικό. Επίσης, ε, αφισβητώ με την έκθεση, με την ε, πρόταση της ε, ε της προέλευσης, γιατί αφαιρεί τον ανθρώπινο παράγοντα. Παρόλο που θεωρώ ότι ο ανθρώπινο παράγοντα είναι πολύ σημαντικό για την έννοια τη προστατευόμενη ονομασία προέλευση. Επίση, τα ο ίνος χωρίς ε, αλκοόλ δεν είναι ίνος κατά τη γνώμη μου. Η νέα κατηγορία δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό που προτείνει η ΚΟΑ. Αντίθετα, ε, είμαι υπέρ ε, αυτών των προϊόντων χωρίς αλκοόλ, αλλά δεν έχουν, δεν έχουν θέση στην ΚΟΑ να μείνουν αλλά όχι στην ΚΟΑ. Επίση, είναι υπέρ τη απλούστευση των διαδικασιών προστασία του συστήματο ποιότητα των ίνων και καλύτερη προστασία για τα κρασιά υπό διαμετακόμιση που πολλούνται μέσω ίντερνετ. Επίσης είμαι κατά των χρήσεων που αποδυναμώνουν τη φήμη των ποιοτικών ίνων και των κακόπιστων εγγραφών ή παρόμοιων τομέων που μπορούν να επηρεάσουν τα ποιοτικά κρασιά. Επίσης θέλω διευρυμένο έλεγχο για να καταπολεμήσουμε κάποιες αμπελονικές απάντες. Και κάτι που δεν αναφέρεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την ετικετοθεσία του κρασιού. Γιατί τίποτα δεν αναφέρεται στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προτείνω μετά από συνεννόηση με τον κλάδο να καταστήσουμε υποχρεωτική την επισήμανση των ίνων και για την θερμιδική του αξία και για, τη, για τον κατάλογο των συστατικών που περιέχουν γιατί η θερμιδική αξία θα πρέπει να αναφέρεται στην ετικέτα του ίνου και επίσης τα συστατικά θα πρέπει κατ' επιλογή του αμπελουργού είτε να αναφέρονται στην ετικέτα είτε να μπορούν να τα βρίσκουν εξ αποστάσεως τα στοιχεία αυτά οι καταναλωτές. Επίσης, για την προθεσμία της εφαρμογής. Το έργο συνεχίζεται, ακόμα είμαστε σε φάση υποβολή σχεδίου έκθεσης. Θα εξελιχθεί φυσικά αυτή η έκθεση και εγώ θα τροποποιήσω την έκθεσή μου γιατί το κρασί είναι ένα ζωντανό προϊόν και η έκθεση επίσης είναι μια δυναμική διαδικασία και πέραν των προτάσεων που έκανα ε, να αναφέρονται οι θερμίδε ε, ε, με βάση κατεξοδότηση πράξη. Εγώ πιστεύω, ανάλογα και με τι απαιτήσει των καταναλωτών, να αναφέρονται οι θερμίδε το χρόνο που ακολουθεί την βασική ε, νομοθετική πράξη. Φαίνεται ότι ο μπελονικό κλάδο δεν είναι κατά αυτή τη πρόταση. Αντίθετα, ίσω θα πρέπει να διαπραγματευτούμε την προθεσμία για τον ορισμό των συστατικών, γιατί από τεχνική άποψη ίσω δημιουργηθούν κάποια προβλήματα στον κλάδο. Δεν θέλουμε να παρεμποδίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου, αλλά να δώσουμε κάποια στοιχεία ε, ε, που θα βοηθήσουν τον καταναλωτή χωρίς να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του αμπελονικού τομέα. Αυτά ως προς τον αμπελονικό τομέα. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ποιότητα. Συμφωνώ με τις προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλούστευση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας και να διευρύνουμε την πολιτική ποιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, είμαι κατά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέλει να καταργήσει από τη συγγραφή υποχρεώσεων των γεωγραφικών ενδείξεων κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν προέρχεται από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι ε, λάθος και κίνδυνος. Για παράδειγμα, ε, για, την για ένα προϊόν που είναι αυτόχθονο, προϊόν της ε, Κορσικής, για παράδειγμα πώς ε, θα δίνεται το πιστοποιητικό κορσικό αλλαντικό αν δεν υπάρχει διαβεβαίωση που προέρχεται από την κορσική αυτό το προϊόν. Αυτό λέω εγώ στην πρότασή μου. Δεν θα πρέπει να καταργείται η γεωγραφική προέλευση του προϊόντος για να μην υπάρχει καμία αφιβολία. Σε ό,τι αφορά τον Ίνο, προτείνω ε, ευθυγράμμιση ε, των ορισμών γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασίας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης με τα όσα αναφέρονται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Σε ό,τι αφορά την γεωργία των εξόχω απόκεντρων περιοχών και των νησιών του Αιγαίου, προτείνω να μειωθούν τα κονδύλια που προτείνονται Ευρωπαϊκή, να μην μειωθούν τα κονδύλια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επανέλθουμε στα αρχικά ποσά. Και ένα άλλο βασικό στοιχείο της πρότασής μου αφορά το θέμα της ρύθμισης. Θα πρέπει εδώ να δούμε ποια είναι τα διακυβευόμενα. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν λαμβάνει σωστά υπόψη την απώλεια εισοδήματο ή την μεγάλη αστάθεια των τιμών. Και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σιώπησε πλήρω ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλο τη κοινή γεωργική πολιτική δεν ε, ανταποκρίνεται στι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Αυτός ο προσανατολισμός ε, είναι ιδεολογικός και τα αφήνει όλα ελεύθερα. Κάτι που δεν ε, ανταποκρίνεται στις δυσκολίες ε, της εποχής αυτής. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα λάθη του παρελθόντο, αλλά θα πρέπει να επιφέρουμε κάποια αριθμιστικά στοιχεία στην κοινή γεωργική πολιτική και να την προσαρμόσουμε, να προσαρμόσουμε του ε, υπάρχοντε μηχανισμού τη ΚΟΑ στι νέε συνθήκε. Και αυτό που προτείνω στην έκθεσή μου είναι να προσθέσουμε έξι επιπλέον μηχανισμούς σε όλους τους τομείς, ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν έγκαιρα ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτοί οι μηχανισμοί ε, κινητοποιούν τις δημόσιες αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επαγγελματικέ οργανώσεις. Και μετά την ανταλλαγή απόψεων ε, που είχαμε με τον κύριο Χόγκαν, θα ήθελα να κάνω μία ε, ερωτική εξομολόγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί στην ερωτική εξομολόγηση δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε ε, λόγια, αλλά θέλουμε και έργα που να αποδεικνύουν τον έρωτα, την αγάπη. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει το ρόλο του τομεακού ρυθμιστή ουσιαστικά. Και αυτό θα ήθελα να εξασφαλίσουμε. Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη και διαχείριση των κρίσεων, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτή είναι η πρότασή μου, να υποβάλει δύο έγγραφα. Ένα που να αφορά τα χαρακτηριστικά τα, τα, των διαφόρων ειδών κρίσεων και πέραν τούτου να μας λέει τι λύσεις θα προτείνει σε περίπτωση κρίσης ανάλογα με τα διάφορα είδη κρίσεων ή προκλήσεων. Αυτό είναι προπετούμενο της πρότασης μου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ορίσει τι εννοεί ως κρίση. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των αγορών. Τα δεδομένα των κρατών μελών, τα δεδομένα των επαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει να διατίθενται για να μπορούμε να καθοδηγήσουμε καλύτερα τις αγορές. Αυτή η διαφάνεια είναι απαραίτητη και μπορεί να μας βοηθήσει και επίσης να μας προειδοποιήσει για κάποιες ε, εισαγωγές με τιμές εισόδου που είναι αρνητικές για την ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης θα μπορούμε να δίνουμε στις ε, εφορίες ε, στοιχεία για τις συναλλαγές ώστε να ελέγξουμε καλύτερα τα παράγωγα γεωργικά προϊόντα. Οπότε θα πρέπει να ορίσουμε στη κρίση. Δεύτερον, να, να βελτιώσουμε την διαφάνεια των αγορών και εκεί θα παίξει ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης να εφαρμόσουμε ένα σύστημα εθελοντικής αποσύρσης της παραγωγής σε περίπτωση κρίσης που θα ισχύει για όλες τις παραγωγές. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της συνεργασίας μεταξύ των τριώθεσμικων οργάνων. Για να μην βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που είχαμε με την κρίση του γάλακτος που περιθωριοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να παραγωνιστούμε, θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε. Και προτείνω κάποια στρατηγικά σημεία σε ένα ιδιαίτερο και συγκεκριμένο πλαίσιο επιδόσεων. Προτείνω λοιπόν αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους φορείς διαχείρισης ε, των κρατών μελών στον πρώτο πυλώνα. Σε ό,τι αφορά το βάρος ε, των παραγωγών στην ε, τροφική αλυσίδα. Μετά την ομολογία για τα γαλλικά και χώρια και το κανονισμό «Ομνιμπος», θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το έργο των συναδέλφων Ταντάν και Ντεκάστρο για τον κανονισμό Omnibus και τη μεγάλη βελτίωση που έγινε. Επίσης θα πρέπει να άρουμε κάποιες αφιβολίες ε, για τους γεωργούς για να επανισορροπήσουμε καλύτερα την ε, δύναμή τους στην ε, αγορά. Σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών, διαγράφουμε τη μνήα στην εκχώρηση ιδιοκτησίας. Και επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε τη ρήτρα των τιμών που δεν είναι πια επίκαιρη. Σε ό,τι αφορά τι διαπαγγελματικέ οργανώσει, δυνατότητα ε, σύναψη τριμερών συμβάσεων για να γίνει κατανομή της αξίας πέραν του πρώτου αγοραστή. Τρίτον, και θα ολοκληρώσω εδώ, το θέμα της δημόσιας παρέμβασης. Προτείνω διεύρυνση και στο χείριο και ε, πρόβιο κρέας και να ληφθεί υπόψη επίσης δημόσια παρέμβαση, το Brexit και τα προβλήματα στην υγεία που δημιουργεί η ε, νόσος, η τελευταία επιζωτία στους χείρους και επίση θα ληφθεί υπόψη ε, την αναπροσαρμογή των τιμών. Προτείνω κάποιους κανόνες για την εμπορευματοποίηση, για το βόλιο, εγωπρόβιο, κρέα, τα γαλακτοκομικά, κάτι που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, προκειμένου να, εμποδι... να εξασφαλίσουμε εμπορία τους, ε, να έχουμε θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ κοινοτικών και εξοκοινοτικών παραγωγών με βάση την αρχή τη αμοιβαιότητα και επίση να ληφθούν υπόψη νέε προσδοκίε των καταναλωτών σε ό,τι αφορά το, το, τι ζωοτροφέ, την ιχνηλασιμότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Τέλο, ό,τι αφορά τη ρυθμίση τη προσφορά, προτείνω να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα που έχουν το σήμα τη ε, εθνική ή ευρωπαϊκή ποιότητα. Γεωγραφικέ ενδείξει, προστατευόμενη ονομασία προέλευση κτλ να μπορούμε να ρυθμίζουμε για αυτές τις ενδείξεις. Και σε ό,τι αφορά τις αγωγές από τρίτες χώρες, θέλουμε μία ρήτρα διασφάλισης για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Αυτά και σας ευχαριστώ που με επιτρέψετε να σας κάνω μία σύνοψη της έκθεσής μου. Παρακαλώ, οι υπόλοιποι αστηρίσουν το χρόνο τους. 1,5 λεπτό το πολύ. Σας θέρμο παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Προσπαθήσω, Πρόεδρο. Η έκθεση του συναδελφού Αντριέ είναι ένας αξιοθαύμαστος όγκος εργασίας και αναλύει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα σημείο και μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά τα οποία προτείνονται για την πολιτική ποιότητα, για τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, για τις πότερες περιφέρειες και για την ε, περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Παρακολουθήσαμε την ε, εξέλιξη όσον αφορά την κοινή οργάνωση της αγοράς, αλλά δεν θα πρέπει να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας όσον αφορά τις ε, εξελίξεις που ε, καταφέραμε να αποσπάσουμε, να εξασφαλίσουμε μέσω του ομνίμπους. Και έχουμε τρεις άξονες εδώ, σταθεροποίηση, διαφάνειες αγορές, στην οργανωσή αγοράς υπάρχουν όλα τα μέσα για εξασφάλιση της διαφάνειας. Ήδη τα είναι και αυτό το κοινοβούλιο το 13 θα ε, πρέπει τώρα όλα αυτά να τα αποσπάσουμε από το Συμβούλιο που είχε πει όχι την τελευταία φορά. Ε, τώρα για την αλυσίδα της προμήθειας τώρα έχουμε την έκθεση Ντεκάστρο βρίσκεται σε φάση τεμέρους διαλόγου θα πρέπει να συμπληρωθεί ό,τι χρειάζεται αλλά όσον αφορά την προστασία των προϊόντων ποιότητας εδώ θα πρέπει να είμαστε ε, κατηγορηματική και να υπάρξει κάποιο είδου αποκέντρωση στην διαδικασία και να πετύχουμε αυτά τα δευτερεύοντα που θέλουμε. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το ότι υπάρχουν κάποια μέσα για τη διαχείριση της αγοράς αλλά θα πρέπει να γίνει η διάκριση από τα μέσα διαχείρισης των μεγάλων ε, κρίσεων. Έχουμε 400 εκατομμύρια. Αυτά είναι για τις σοβαρές κρίσεις. Δεν είναι για την ε, τακτή διαχείριση της ε, αγοράς. Εδώ έχουμε τη μεγάλη μας διαφορά από την Κομισιόν. Δεν θέλει το ίδιο με μας η Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο θέλει να υπάρξει μια ελάχιστη ρύθμιση. Θα πρέπει αυτά να είναι κατανοητά και έτσι να υπάρξει εμπιστοσύνη στην αγορά. δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε την εξασφάλιση των ε, γεωργών μας. Και προσοχή να μην έχουμε εμεί τα δρακόντια μέτρα και όχι ο υπόλοιπο κόσμο. Πρόεδρος. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ανδριό για την έκθεσή του, για την πλήρη έκθεσή του, για το Omnibus Είμαστε ούτω ή άλλως ε, πολύ ε, ενεργοί στη συμμετοχή μας και για την ΚΟΑ. Ε, νομίζω ότι πλέον δεν έχουμε πολλά να κάνουμε. Οι προτάσεις πλέον είναι επιτάπητο και θα τις μελετήσουμε πολύ προσεκτικά. Οι προτάσεις της Κομισιόν για τις γεωγραφικές ενδείξεις νομίζω ότι είναι πολύ θετικές και η απλούστευση του συστήματος με την πιο γρήγορη καταχώρηση και την πιο αποτελεσματική αδειοδότηση για τις αλλαγές των ενδείξεων νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη αλλαγή. Μετά, το, ε, τα προϊόντα ίνου και τον ίνο χωρίς αλκοόλ ε, νομίζω ότι αυτό ανήκει κυρίως ε, ε, στο, στην αίσθηση που μας δημιουργούν τα, ε, τα ποτά αυτά. Ο κυρίως όταν είμαστε με μια παρέα και ή στο δρόμο και θέλουμε να πιούμε ένα κρασί χωρίς αλκοόλ, πάντα ένα ποτήρι κρασί μας δημιουργεί καλύτερα αισθήματα από ότι ένα ποτήρι νερό. Βεβαίω εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν το αλκοόλ, υπάρχουν οι έγκυε γυναίκε. Όλα αυτά όμω θα τα λάβουμε υπόψη. Κατά την άποψή μου, Εν τω μεταξύ υπάρχει τόσο πολύ ε, τόσο πολύς έλεγχος και έρευνα που δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαγορεύουμε ποικιλίε και για, το, για τις οργανώσεις παραγωγών για το γάλα θα πρέπει να σκεφτούμε αν χρειαζόμαστε αριθμητικά στοιχεία ή αν πρέπει να πούμε ότι οι οργανώσεις αγορών θα βρίσκονται στις, στους ίδιους, θα πληρούν τους ίδιους όρους με τους ε, γαλακτοπαραγωγούς. Ευχαριστώ. Βάιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συνάδελφο Αντριώ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Εφόσον πρέπει να κάνουμε παρεμβάσει στην αγορά, νομίζω ότι έχουμε την ε, ε, κατάλληλη χρονική στιγμή για να τι εποπτεύσουμε κιόλα. Με είναι εποπτική αυτή δυνατότητα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιε είναι οι παρεμβάσει που χρειάζονται και να έχουμε καλύτερου μηχανισμού. Οπότε τέτοιου είδου παρεμβάσει θα κάνουμε εμεί. Είναι πραγματικά σημαντικό το εργαλείο αυτό, το μέσο αυτό και θα πρέπει ίσω να σκεφτούμε μήπω οι οργανώσει παραγωγών να ε, τη συμπεριλάβουμε ανά ε, είδος παραγωγής, ας πούμε βιολογική παραγωγή και όχι ένα προϊόν. Για τα είδη τώρα του κρασιού, συμφωνώ με τη συναδελφό Μίλλερ. Εδώ θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ποικιλίε να επιτρέπονται σε ό,τι αφορά και την, αγορά, και την αλλαγή στο κλίμα και την ε, λυπή χρήση ζενιοκτώνων και για την επισήμανση θα πρέπει να υπάρχει, να γίνεται παραπομπή σε μία ιστοσελίδα και εκεί να διατίθενται όλα τα δεδομένα, γιατί αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για, την, για τους μικρούς παραγωγούς. E Ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριε εισηγητά. Πολλά είναι τα θέματα που αναφέρθηκαν. Στα πιο σημαντικά θα επικεντρωθώ. Οι διατάξει όσον αφορά τον έλεγχο της προσφοράς. Είναι η επιλογή ευφυής, οπότε συμφωνούμε όσον αφορά το ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τη χρήση των εύρυθμα των μηχανισμών από άλλους κλάδους. Επίσης, καλό είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία ε, και έτσι να υπάρχουν θεμητές ε, να είναι θεμητός συντονισμός και όσον αφορά αυτό το ε, τομέα θα πρέπει να δούμε ε, τι αλλαγές έχουν γίνει όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης ε, και να έχουμε υπόψη τη συμφωνία TRIPS. Ο άνθρωπος παράγων είναι απαραίτητο στην προσφορά του και εκεί θα πρέπει το βάρος τόσο. Και Εμάς μας ανησυχεί το ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποια ε, είδη που μέχρι τώρα δεν επιτρεπόντουσαν. Να μην υποτιμούμε τις παραδοσιακέ ποικιλίε. Να μην έχουμε την προσφυγή σε εισαγωγές από τρίτες χώρες εκεί όπου ήδη καλλιεργούνται αυτές οι ποικιλίε. Τώρα γιατί την σε αλκοόλ ε, θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την παράδοσή μας. Είναι περισσότερο βιομηχανικά προϊόντα. Ευχαριστώ κύριε Σκολομπία. Ευχαριστώ. Η έκθεση του συναδέλφου Αντριέ περιλαμβάνει κάποιες ε, εύστοχες παρατηρήσεις αλλά και μερικές άστοχες. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ε, μιας κατηγορίας κρασιού χωρίς αλκοόλ ή των ε, κατηγοριών χωρίς αλκοόλ που δεν ανταποκρίνεται στο, στο παράρτημα 7.2 του ΚΟΑ γιατί τα κρασιά αυτά χωρίς αλκοόλ ε, χρήζουν ε, κάποιων αρωματικών ουσιών και άρα στην κατηγορία των βιομηχανικών προϊόντων. Επίπτουν στον κανονισμό 251 του 2014 για το αρωματισμένα κρασιά. Ε, περισσότερο μοιάζουν με χυμούς φρούτων παρά με ίνους. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την επέκταση στη ζάχαρη και στο χείριο κρέας των Ατσικόα. Ε, και για τις πιθανότητες ε, ταραχής που θα έχει, διαταραχής των αγορών που θα έχει το Brexit μετά την ε, ε, επιζωτία για τους χείρους. Επίσης, μετά την απελευθέρωση των ποσοστώσεων είχαμε αύξηση της τιμής και παρόλα την παταγώδη αποτυχία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει παρέμβει στην αγορά και είναι υπέρ της απορρίθμισης. Αυτές οι τρεις παραγωγέ θα μπορούσαν να υποφεληθούν από την ιδιωτική αποθεματοποίηση και προτείνουμε να περιληφθούν στο κατάλογο των προϊόντων που θα μπορούσαν να περιληφθούν στη δημόσια παρέμβαση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έρντος. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σύντομα να σας αναφέρω μόνο δύο συγκεκριμένα θέματα για τα οποία σας ακούσαμε. θα πρέπει να μην έχουμε περικοπές στους πόρους. Θα πρέπει να υπάρχει ρύθμιση μια αναλογικότητα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για την κοινή οργάνωση αγοράς. όπως είπαμε και για την έκθεση Εράθ Γκαρθία. Επίσης, προσοχή να μην κάνουμε κινήσεις που λιμονούν κινδύνους για την παραγωγή του ίνου. Να υπάρχει πρόσταση γεωγραφικής προέλευσης και να προστατεύσουμε την ποιότητα του ίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρει παρατηρήσει σύντομα για το κρασί, για τον ίνο. Για την. Για την ε, σύμπτυξη των ε, ε, ποικιλιών θα πρέπει νομίζω να την επιτρέψουμε όπως είχαμε πει. Βεβαίως για κάποια σημεία θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως ε, έχουμε 5.000 διαφορετικές ποικιλίε ε, σταφυλιών στην ε, Ευρώπη. Έχουμε και την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να είμαστε σίγουροι να μην... δεν κάνουμε χάρη στην ποιότητα του κρασιού της Ευρώπης. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε περισσότερες απαιτήσει. Τώρα για το κρασί χωρίς αλκοόλ, αφού μπορούμε να προσθέσουμε είτε αλκοόλ είτε ζάχαρη, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Τι γίνεται με την πύρα, αν πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μία μπύρα ε, ή ένα ποτό χωρίς αλκοόλ που βασίζεται στην πύρα. Ε, αστεία πράγματα τώρα, δεν είναι αυτά. Νομίζω ότι ε, και για το κρασί κάτι α, ανάλογα πρέπει να κάνουμε. Εγώ είμαι και εισηγητής για την ε, γνωμοδότηση αυτή στην ΕΝΒΗ ο εισηγητής Αντριέ αλλάζει με την έκθεση του τους κανόνες για την επισήμανση. Αυτό δεν είναι όμως αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Η επισήμανση των, τροφών, των τροφίμων είναι αρμοδιότητα της ΕΜΒΗ. Οπότε την... είναι σαν να προσπαθούσε η ΕΜΒΗ να αλλάξει την ε, κοινή αγροτική πολιτική. Καταλαβαίνετε. 53 συν. Ούτω ή άλλω το έχουμε δουλέψει στην ΕΝΒ. Εγώ δεν έχω επαφή βέβαια με τον εισηγητή. Από ό,τι ξέρω, υπήρξε στην Άγκρη μια σκιώδη συνάντηση όπου δεν με προσκάλεσε κανεί και έγιναν κάποιε ανταλλαγέ απόψεων τέλο πάντων μεταξύ των εκπροσώπων των δύο επιτροπών. Καλό θα ήταν να μείνουμε ο καθένα στι αρμοδιότητέ μα, ωστόσο. Εμεί επιμένουμε στι δικέ μα. Ε, υπάρχουν θέματα που είναι ευαίσθητα για του ε, συναδέλφου, αλλά νομίζω ότι δεν ε, θα καταλήξουμε κάπου αν προχωρήσουμε έτσι. Οπότε παρακαλώ να αλλάξει λίγο την προσέγγιση του ο εισηγητή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις, τις αρμοδιότητες των Επιτροπών. Σα παρακαλώ, να τηρείτε το χρόνο σα, αλλιώ δεν θα προφτάσουμε. Κυρία Ντελαγία. Πολύ σύντομη θα είμαι γιατί με κάλυψαν οι προλαλήσαντε. Για τη διεύρυνση του καταλόγου για τα προϊόντα, αναφερθήκατε στο χείριο και στο πρόβιο να περιληφθεί και η ζάχαρη. Επίσης, ε, πατείται μείωση του προπολογισμού για τις εξόχως απόκεντρες και τις νησιωτικές περιοχές. Ε, Ζητούμε επαναφορά των κονδυλίων. Επίσης, ε, να προσέξουμε τα θέματα του ίνου σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις παραγωγών. Είμαστε υπέρ των βραχαίων αλυσίδων προμήθειας και αυτό ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών. Αυτή του την θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη στη ΣΚΟΑ. Κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ. Ένα σημείο μόνο. Αυτή η στρατηγική του εισηγητού για τις κρίσεις στην αγορά να υπάρχει μια δυνατότητα διαχείρισης κατά τη διάρκεια κρίσεις, ε, με θελοντικές μειώσεις. Ε, ε, νομίζω μάθαμε το μαθημά μας από την κρίση στο γάλα Μειώθηκαν οι τιμέ για το γάλα, πολλέ επιδοτήσει ε, τελικά πετάχτηκαν έξω το παράθυρο. Ε, θέλουμε να υπάρχει ένα μηχανισμό. έχουμε και, έναν, ε, και μια υποπτική αρχή, έναν υποπτικό φορέα, ο οποίο όμω ο φορέα πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί όντω να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου κρίσεις και από αυτού πρέπει να επιμείνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θυμίζω και την σχετική γνωμοδότηση τη οποία ήμουνα η συγγήτρια για την υπερπαραγωγή που ε, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές των αναπτυσσόμενων ε, χωρών. Ε, νομίζω ότι εδώ πρέπει λιγάκι να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά. Ο κύριος Τεσάντος. Δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο της πρότασης. Στα ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομική βάση που αναγνωρίζει τις ε, ιδιαίτερες προκλήσεις αυτών των εξόχων, εξόχων απόκεντρων προϊόχων. Το 2016 έγινε μια αξιολόγηση του ΠΟΖΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ιδιαιτερότητε αυτών των περιοχών δεν καλύπτονται από τα τρέχοντα μέτρα του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ. Οπότε είναι αναφυσβήτητο τη ανάγκη διατήρησης ε, του καθεστώτος αυτού, του προγράμματος και φυσικά με την ε, δέουσα χρηματοδότηση για το ΠΟΖΕΙ. Ε, ζητώ λοιπόν την υποστήριξή σας και όπως πρότεινε ο Ερικ Αντριέ θα ήθελα να απορρίψουμε την περικοπή των δαπανών που προτείνει για το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούμε επαναφορά και ενίσχυση μάλλον των κονδυλίων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και να καλύψουμε τις ελλείψεις που δημιουργήθηκαν λόγω της περικοπής. Αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ. Εράς Γκαρσία. Τέσσερα σχόλια. Ε, φυσικά να διατηρήσουμε τα κονδύλια του Ποσέη. Σε ό,τι αφορά την... Δεν ακούγεστε καλά, κυρία Γκαρσία. Ε, είναι παρακινδυνευμένο αυτό τις προθεσμίες του 2030 για τις εγκρίσει, γιατί προτείνεται να αναθεώρηση το 2023. Καλύτερα να μιλήσουμε για ολοκλήρωση το 2040-2050, γιατί συμφωνώ με την πρόθεση, αλλά δεν ξέρω αν αυτή η πρόταση για το 2023. Σε ό,τι αφορά το, την ποικιλία Λαμπρούσκα, δεν ξέρω αν μια ευρυδική ποικιλία για ε, ίνος με γεωγραφική ένδειξη και pop ε, χαρακτηρίζεται από ποιότητα. Ίσα ίσα αυτός, αυτό το κρασί δεν είναι και πολύ καλής ποιότητας. Έχουμε μια υβριδική ποικιλία που δεν ανταποκρίνεται στις ψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Συμφωνώ με τη διαγραφή του άρθρου 222. Ε, Θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα αυτό στο, στις διαπαγγελματικές οργανώσεις ε, διαφωνώ με τη διαγραφή μάλλον. Ίσως να τροποποιήσουμε το μηχανισμό, αλλά όχι να το διαγράψουμε πλήρως. Κυρία Ριμπέιρο, ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί ενδιαφέρεται για τη χρηματοδότηση του ΠΟΖΕΙ. Πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε το ΠΟΖΕΙ. Ο ίδιος ο Επίτροπος Χόγκαρ όταν πήγε στις Αζόρες μετά από δική μου πρόσκληση τον περασμένο Ιούνιο είπε ότι δεν θα μειώσει τη χρηματοδότηση του ΠΟΖΕΙ. Θα πρέπει σε αυτό να είμαστε αδιάλακτοι και ανένδοτοι. Να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός του ΠΟΖΕΙ για να μην έχουμε συνέχεια προβλήματα στι διαπραγματεύσει. Επίσης, σύντομα θα ήθελα να αφαιρθώ στην ανάγκη τη αυτονομίας του ΠΟΖΕΙ και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Και μάλιστα έχω καταθέσει σχετικέ ε, τροπολογίε. Για τον πρώτο πυλώνα, το ΠΟΖΕΙ δεν μπορεί να εξαρτάται από τα στρατηγικά σχέδια τη ΚΑΠ. Και σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη, δεν μπορούμε να έχουμε ε, την κεντρική κυβέρνηση να να επεμβαίνει ως διαμεσολαβητής σε μια διαπραγμάτευση που θα πρέπει καταρχήν να είναι άμεση μεταξύ των περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Δεκάστρο. Σύντομα, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα, Ερίκα για την πολύ καλή δουλειά σε τόσο σύντομο χρόνο. Η έκθεση αυτή είναι σημαντική βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν σε πολλά σημεία για την ποιότητα της ε, και ενδύσεις, για, τα, για τη διαχείριση της ε, προσφοράς ε, σε σχέση με την προηγούμενη ΚΑΠ, για τη διαφάνεια της ε, αγοράς, όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με τη δουλειά που κάνουμε στον με τις πρακτικές. Ο ΕΡΙΚ έχει φιλόδοξες ιδέες όσον αφορά τον ανταγωνισμό, οπότε παρόλα αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Μισελ Νταντέν θα πρέπει να μετέλθουμε του, του, και να μην ξανανοίξουμε εκείνη την τόσο δύσκολη προβληματική που θυμίζω ότι είχαμε ολοκληρώσει με αυτήν την ε, σημείωση στο περιθώριο. Προσοχή, προσοχή εδώ, αυτό σας επισημαίνω. Κατά τα λοιπά, συμφωνούμε με τον ε, Ερικ. Κύριε Καπούτο. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Ρίκ και γιατί ανέβασε τον πύχη σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε συμφωνώ με όλα όσα προτείνει. Να συνεχιστεί η κρατική παρέμβαση, να υπάρξει αυτό το δίκτυο ασφαλείας από δεν υπάρχει άλλο μέσον, να αναβαθμιστεί ο ρόλο των μέσων των παραγωγών. Όπω είπε και ο Ερικ, να χρησιμοποιήσουμε τι νέε τεχνολογίε πληροφορική για επικοινωνίε, τα blockchain και έτσι να απλουστευτεί η δουλειά στην καλλιέργεια και στην ε, διανομή των προϊόντων για τα αμπελοϊνικά. Ε, συμφωνώ 100% ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις για τη φύτευση και με κατά, όπως και έριξε την πρόταση της Κομισιόν που θέλει να αλλάξει τον ορισμό ε, της προστασίας εν, των ενδείξεων. Τώρα όσον αφορά τα κρασιά χωρίς ε, αλκοόλ, ναι, να δούμε τη στάση της αγοράς. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει η διάκριση σε σχέση με το κανονικό κρασί και τόσο προβλέπει η κοινή οργάνωση αγοράς. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας τονίσατε το ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτήν την ε, σύντομη αλυσίδα προσφοράς. Να υπάρχει μια αγορά όπου να μπορεί ο Γιωργός να θέσει συμπορία τα προϊόντα του. Περνάνε τώρα μεγάλες δυσκολίες. Θα πρέπει να οθυγούμε ο ορισμός αυτής της ε, αλυσίδας προσφοράς. Θα τους βοηθούσε. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε μέσα σε πέντε λεπτά κύριε Μέγκελε να μας δώσετε απαντήσεις. Θα ήμουν... Πρόεδρε ευχαριστώ να είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί σε 6.30 έχω ένα τριμερή διάλογο με περιμένουν γιατί και εκεί έχουμε σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Μας παρουσίασε μια πολύ μεστή έκθεση από ιδέες. Αν το κάναμε σε αυτό, χρειαζόταν επί 1,5 χρόνο να δουλεύουμε για τη μελέτη των επιπτώσεων. Και γι' αυτό και διαλέξαμε κάτι φτωχότερο λιτότερο. Σωστό είναι το ότι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αρκετά είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της έκθεσης και του κανονισμού της οργάνωσης αγοράς και άλλων κανονισμών. Και ένα σημείο επίσης το οποίο μας διέφυγε τελείως όλων είναι η πρόταση του κανονισμού στρατηγικού σχεδίου το να ξεκινήσουμε κάποια λειτουργικά προγράμματα για τι οργανώσει παραγών σε άλλου τομεί. Αυτό το 3% του προπολογισμού που προβλέπεται για τέτοια μέτρα που θα έχουν ε, σημαντική επιρροή όσον αφορά την διαχείριση της, του ιδιωτικού τομέα στην αγορά. Τι γίνεται επίσης με την αλυσίδα της προσφοράς, των διατροφής, θα πρέπει να δούμε ότι είναι πολύ σημαντική συνέπεια μεταξύ των πολιτικών. Να το δούμε. Δύο λόγια το για, αυτή την διατροφική αλυσίδα και την αγορά. Για τη διαχείριση της αγοράς εμείς διστάσαμε να προτείνουμε κάτι. Γιατί θεωρούμε ότι η πολιτική απόχωρηση που υπήρχε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει προστολισμός προς την αγορά. Να είναι εύρεθμη η λειτουργία επίσης του δικτύου ασφαλείας. Και τώρα, ο εισηγητής πάει ακόμα παραπέρα από το δίκτυο ασφαλείας. Το θέμα είναι τώρα αυτό τι θα είναι. Παρέκκληση ή μια πλήρης στροφή κατεύθυνσης της ΚΑΠ να μην έχει πια προσανατολισμό της αγοράς. Τα το συνέδριο για τις άμεσες πληρωμές. Αν τα μέτρα για την αγορά έχουν ακόμα περισσότερες επιπτώσεις, ε, τότε τι θα γίνει με τις άμεσες πληρωμές, τις ε, συνδεόμενες πληρωμές, συνδεδεμένες τέλος πάντων, θα πρέπει και αυτές να αυξηθούν αντίστοιχα. Τι γίνεται τώρα με την αριθμική προσαρμογή. Ε, εδώ τότε απαιτείται παρέμβαση με δημοσιονομικές συνέπειες. Και το είναι πού θα πάνε τα προϊόντα όταν φύγουν από την αποθεματοποίηση. Τι γίνεται. Είδατε τι έγινε με το γάλα σε σκόνη, το αποβιτηρωμένο. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα απόσυρσης που θεσπίσαμε κατά την κρίση του γάλακτος για όλους τους κλάδους. Και κάπως με ενοχλεί το ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να δούμε το τι μήνυμα θα στείλουμε με αυτά τα μέτρα προς τους παραγωγούς. Τώρα, τα μέτρα για την κρίση το του με τον οριζόντιο διαγωνισμό. προσπάθησα να σας εξηγήσω την προσέγγιση μας. Σίγουρα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η διάρκεια μεταξύ μέτρων κρίσης και μέτρων αγοράς. Αλλά βέβαια, πάντα το ερώτημα είναι από πού θα βγουν τα λεφτά. Αν είναι από τον προϋπολογισμό, αυτό είναι το πιο εύκολο, το πιο πρακτικό, ούτως ώστε να έχουμε το αποθεματικό αυτό. Και τώρα για την διατροφική αλυσίδα, σας παραπέμπω σε όσο είπε ο κύριο Νταντέν. Πολλά πετύχαμε με το Omnibus πριν από ένα χρόνο. Τι να κάνουμε, να ξανοίξουν το κουτί της Πανδώρας μετά το όσο πετύχαμε. Καλά το είπατε κύριε Νταντέν. Θα θέσουμε κινδύνο όλα μας τα επιτεύγματα για τη διαφανεία στην αγορά θα ξέρετε ότι τώρα προβαίνουμε σε κάποια ενδελεχή ανάλυση. Στη συνέχεια θα έχουμε νέα μέτρα για περισσότερη διαφάνεια στις τιμές που αφορούν την διατροφική αλυσίδα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα για το δίκαιο ανταγωνισμό έχουμε ένα νέο νομοθέτημα θα πρέπει να δοκιμαστεί και μετά να δούμε αν θέλει αναθεώρηση. Για να δούμε τώρα τη δέσμη μέτρων για το κρασί. Μας λέει ο συγκητή ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα αδειοδότηση παράταση μετά το 2030, χωρίς όριο. Είπαμε τα σχετικά με τα δικαιώματα φύτευσης και το 2030 και μετά από έχουν γίνει είπαμε να υπάρχει παγίωση του προγράμματος και να γίνει ένα πρόγραμμα αξιολόγησης για το 23. Αν τότε όμως δεν χρειάζεται να υπάρχει τέτοια αξιολόγηση εάν ε, συμφωνήσουμε για μια αυτή παράταση χωρίς τέλος, χωρίς τέρμα και βλέπω και χαίρομαι που συμφωνεί ο εισηγητής ότι Θέλουμε να σταματήσει η απαγόρευση σχετική με τις απαγορευμένες ποικιλίε. Τα κρατη να χαρακτηρίσουν, να κατηγοριοποιήσουν κάπου τα βήτης λαμπρούσκα, αυτές τις ποικιλίε ή την ποικιλία. Ε, δεν υπάρχει πια αιτία για απαγόρευση από τη βάση του περιβάλλοντος ή της ε, υγείας. Τώρα τα κανονικά γρασιά και τα άλλα, τα, τα μία αλκοολούχα κλπ. Αν θα πρέπει να εξισώνονται όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Το θέμα τι θα γίνει στην αυριανή αγορά. Περισσότερο συνταγωνισμό, περισσότερη παγκοσμιοποίηση στην αγορά. Και άρα θα πρέπει η πολιτική μα να αποσκοπεί στον έχουν όλα τα μέσα οι οποίοι ούτω ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα να προστατεύουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κρασιού και στο μέλλον κάθε κρασί χωρίς ε, αλκοόλ θα προέρχεται από το κρασί. Άρα γιατί να θεσπίσουμε κάτι που θα θεωρείται νέο και δεν θα προέρχεται από κρασί. Καλύπτει το θέμα της ετικετοθεσίας, των διατροφικών χαρακτηριστικών. Αυτά όλα είναι στον κανονισμό 1308 και άρα θα πρέπει να συζητήσουμε ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη τα όσα θέλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου. Η πρότασή μας του 2018 δεν υπήρχε πρόταση για άλλα υποχρεωτικά στοιχεία όπως προβλέπει ο 1308 γιατί έχουμε την έκθεση του 2017 της Επιτροπής για την υποχρεωτική ετικετοθεσία για τα διατροφικά χαρακτηριστικά και επίσης υπάρχει νομοθεσία για την βιομηχανία αναψυκτικών. Ο δε κλάδος είναι υπέρ της πρότασής μας για τα κρασιά ιδίω μετά από τα προβλήματα της αυτορύθμισης και είχαμε και πρωτοβουλίες κρατών μόνο για την ετικετοθεσία που θα μπορούσε να υπάρχει κίνδυνος για τη λειτουργία της ε, ενίας αγοράς. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και θα ακολουθήσουμε τις εξελίξεις τώρα όσον αφορά to improve our γεωγραφικές ενδείξεις. Όποτε θέλετε να τα συζητήσουμε. Έχουμε πνεύμα διάθεση συζήτηση. Εδώ θα βάλουμε τελεία και βέβαια όπως πάντα Ό,τι θέλετε σε τεχνικό επίπεδο να το συζητήσουμε. Να σας εξηγήσουμε την πρότασή μας και να σας εξηγήσουμε. Γιατί επιφυλασσόμαστε για κάποια σημεία που περιέχονται στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Αντρία. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να απαντήσω όλα όσα ακούσαμε. Και μπορώ, θα μπορούσα ανάποδα να ξεκινήσω από αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν συμφωνώ με την Επιτροπή όλα καλά. Με το που αφισβητούμε κάτι αρχίζει και στραβώνει το θέμα. Και φυσικά είναι σημαντικό το θέμα του αμπελονικού κλάδου αλλά εδώ έχουμε μόνο 3%. Ενώ όταν έχουμε μεγάλο κλάδο όπως του κρέατος, τότε το πρόβλημα διευρύνεται. Και αν έχουμε μόνο μία κόα στο ενιαία, πιστεύω ότι θα καταναλώσει το σύνολο του κονδυλίου. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις, οπότε ξέρω αν τα μέσα θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε όλους τους τομείς. Πάντω για να καθησυχάσω τον κύριο Νταντά, τον Παόλο Ντεκάστρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι φυσικά δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε σε σχέση με τα επιτεύγματα του Omnibus. Ούτε θέλουμε παλινδρόμηση σε σχέση με αυτά που έχουμε επιτύχει. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε περαιτέρω, να προοδεύσουμε σε σχέση με τη βάση που δημιουργήσαμε με το Omnibus. Τώρα, αν είναι πολύ νωρί ή πολύ αργά, Προσοχή όμως, ε, όχι να αλλάζουν τα χαόλα και τελικά να μην αλλάζει τίποτα στην ουσία. Θέλουμε να επιταχύνουμε τις εργασίες για ορισμένα θέματα. Σε ό,τι αφορά τα μη αλκοολοχά ποτά, προσοχή, αυτό προτείνει η έκθεση. Δεν είναι ε, να είμαστε κατά των προϊόντων που γίνονται με βάση το κρασί, αλλά χωρίς αλκοόλ εκεί έχουμε βιομηχανικά ουσιαστικά προϊόντα, δηλαδή αρωματικά ουσίνους περισσότερο. Θέλουμε να τα βγάλουμε από την ΚΟΑ όμως αυτά τα προϊόντα, τα μη αλκοόλογα κρασιά. Γιατί αν μπουν στην ΚΟΑ ε, θα λάβουν κάποια κονδύλια και δεν θέλουμε ε, τα κονδύλια της ΚΟΑ να ωφελήσουν άλλο κλάδο πριν του, πλην του αμπελονικού. Και έχουμε το 8,5% ε, αλκοόλ. Αυτό είναι το όριο, για να μην υπάρχει αφησιμία. Δεν θέλουμε να απορρίψουμε αυτό το τμήμα τη αγοράς, αλλά να μην τα χαρακτηρίσουμε ίνο, για να μην ενταχθούν στην ΚΟΑ. Σε ό,τι αφορά τι ποικιλίε. η εισαγωγή νέων ποικιλιών είναι εθελοντική για τα κράτη-μέλη και για τους εμπελουργούς. Υπάρχει δικαίωμα επιλογή Και μάλιστα η μεταρρύθμιση που θα προτείνουμε για την περίοδο 2021-2027 ε, θα πρέπει να προλαμβάνει κάποιες σε ό,τι αφορά τις κλιματικές αλλαγές και τη βιοπικιλότητα. Θέλουμε λοιπόν με την δυνατότητα που προβλέπετε, δυνατότητα όχι υποχρέωση, να χρησιμοποιηθούν νέε ποικιλίε, να καλύψουμε το θέμα της βιοπικιλότητας και να ανταποκριθούμε στι κλιματικέ αλλαγέ ή τη χρήση των λοιπασμάτων στην ε, αμπελουργία. Τίποτα υποχρεωτικό δεν υπάρχει, είναι θελοντική δυνατότητα, προαιρετική. Επίσης, στην έκθεσή μου, ε, που δεν είδε δέχομαι για το ΠΟΣΕΙ περικοπή των κονδυλίων. Και κύριε Ντόρφμαν, για την ειδικατοθεσία ε, δεν συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο την τελευταία φορά. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε όμως για να καθορίσουμε τις αρμοδιότητες μεταξύ των Επιτροπών Έμβη και άγρι. Πάντως, στη μεταρρυθμίση καλό θα είναι να το πούμε. Γιατί έτσι θα το θεσμοθετήσουμε και θα μπορέσουμε καλύτερα να συμπαρασταθούμε στον κλάδο. Δεν πιστεύω ότι είναι ούτε πολύ νωρί ούτε πολύ αργά. Είναι θέμα επίκαιρο και ανταποκρινόμαστε στι απαιτήσει των καταναλωτών αλλά και στη βούληση του κλάδου που είναι αρκετά προοδευτικό. Και μάλιστα ευχαριστώ τους τον ευρωπαϊκό αμπελονικό κλάδο που ασχολήθηκε πολύ με το θέμα και συμφωνεί με την ανάγκη να αναφέρεται η θερμιδική αξία που ανταποκρίνεται σε απέτηση των καταναλωτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέματα των συστατικών, προσθετικών και άλλων ουσιών, αυτό είναι πιο τεχνικό, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα μπορέσουμε να το λύσουμε, γιατί υπάρχει συλλογική βούληση για κάτι τέτοιο. Πάντως ο πελλονικός ε, ευρωπαϊκός τομέας είναι παρόν και στην παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δυναμική των άλλων υπήρων στα θέματα αυτά. Δεν θα πρέπει να φέρουμε σε δυσμενή θέση τον ευρωπαϊκό αμπελονικό τομέα, ούτε να μείνει πίσω σε σχέση με άλλες υπήρους. Και μην ξεχνάτε ότι οι καταναλωτές είναι όλοι και πιο απαιτητικοί ως προς αυτά που καταναλώνουν και τα κρασιά συμπεριλαμβάνονται και σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό θα πρέπει και στις δικές μας προτάσεις να βρούμε αυτές τις ισορροπίες. Αυτά και σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε και περιμένω και εγώ με ανυπομονησία τις τροπολογίες σας για να μπορέσουμε επιγόντως να ξεκινήσουμε τις εργασίες για αυτό το θέμα, την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Τι να πω, να υπενθυμίσω ότι μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου στις μία το μεσημέρι μπορείτε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας όπως και για τις υπόλοιπες νομοθετικές εκθέσεις. Ευχαριστώ, λυπάμαι που σας ε, ζόρισα λίγο και επιταχύναμε, αλλά είχαμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ στο μεταξύ την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, την κυρία Τεκάπελε. Και περνάμε στα σημεία 10 και 11 που προβλέπουν κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Άγκρη και Ντέβε. Το 9 ίσως το συμπεριλάβουμε στην κοινή αυτή συνεδρίαση και μια και που πρέπει να φύγει ο κύριος Δεκάστρο θα ήθελα να μου επιτρέψετε κυρία Δεκάπελεν Πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Δεκάστρο που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Σύνοδο της Μαδρίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μια έκθεση της αποστολής, ε, ε, πολύ κατατοπιστική, ε, που την εκπώνησαν οι γραμματείες της Άγκρη και της ΔΕΒΕ για την κοινή αποστολή στη Μαδρίτη. Είμαστε ο υποφαινόμενος, η Μαρία Χόιμπουχ, η Κλάρα Αγγιλέρα και συνάδελφοι από άλλες επιτροπές, φυσικά και από την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Πολύ σημαντική αυτή η ε, αποστολή. Δεν θέλω ε, να, να μακρηγορήσω τώρα παρουσιάζοντα την πλούσια και με στη μέρα που είχαμε και στη Μαδρίτη. Πάντως η έκθεση της αποστολής αντικατοπτρίζει πιστά τις συζητήσεις που έγιναν στη Μαδρίτη στην Παγκόσμια Κοινοβουλευτική Σύνοδο με την οργάνωση της ε, ε, Ισπανικής Γερουσίας και μάλιστα η ΦΑΟ ε, υπέβαλε κάποια πολύ ανησυχητικά μηνύματα στην συνεδρίαση αυτή και ως επικεφαλής αντιπροσωπείας θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η τήρηση των ε, στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που δυστυχώς φαίνεται όλο και πιο απίθανη όσο προχωρά ο χρόνος. Αυτά όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες τους, πα, παραπέμπω στην λεπτομεριακή έκθεση της αποστολής μας. Σίγουρα είναι τόσο σημαντική έκθεση που πραγματικά θα άξιζε πιο εκτεταμένη συζήτηση, αλλά όχι σήμερα, όχι μια μέρα που μιλήσαμε για τη μεταρρύθμιση όχι μια μέρα που έχουμε τόσο κατάμεστο πρόγραμμα εργασίας. Μια άλλη στιγμή όμως καλό θα ήταν να προβλέψουμε συζήτηση για το θέμα αυτό, γιατί η καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο ε, είναι ένας αγώνας που δυστυχώς ε, πάει προς τα πίσω αντί να προοδεύει. Και νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, γιατί έχουμε αρχίσει και ακολουθούμε μια αρνητική πόρια για την καταπολέμηση της πείνας. Ευχαριστώ. Και η κυρία Χόιμπουχ ήταν μέλος της και αν θέλει το λόγο, ε, μπορεί να μας κάνει μια σύντομη δήλωση. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Παόλο Δικάστρο. Για, αν θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της πείνας παγκοσμίω, πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση είναι δραματική και αυτά που είδαμε στην πρώτη κοινοβουλευτική συνάντηση στη Μαδρίτη θα πρέπει να, την, τα συνεχίσουμε. Οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση. Βεβαίω πρέπει να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε και νομίζω ότι περισσότεροι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να εμπλακούν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό κάποιε χώρε, πόσο λίγε χώρε να, να εκπροσωπούνται στην διάσκεψη αυτή. Η Γερμανία δεν ήταν καν παρούσα. νομίζω λοιπόν ότι πρέπει πιο στοχευμένα να εργαστούμε γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το θέμα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε μια μικρή ενημέρωση, έχουμε λάβει την έκθεση της αντιπροσωπείας και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και ίσως θα έχουμε κάποια ευκαιρία πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας να εγγύψουμε και πάλι σε κοινή συνεδρίαση οι δύο επιτροπές σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Γιατί πολλοί κατηγορούν την ΚΑΠ ότι δεν συμβάλλει αρκετά στην καταπολέμηση της, της πείνας και του υποσυτισμού στον κόσμο. τώρα το 10 το τελειώσαμε. Θα Διεκπαιρεώσουμε τώρα το 11 που είναι στο πλαίσιο της κοινή συνεδρία Άγκρι και στο τέλος θα μιλήσουμε για το 9. Ζητώ συγγνώμη από τους καλεσμένους μας που ήρθαν στο μεταξύ. Θα Έχουμε τώρα την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τόμ Άρνολτ, πρόεδρο τη Ειδική Ομάδα για την Αγροτική Αφρική, σχετικά με το έργο τη Ειδική αυτή Ομάδα. Ας έρθει παρακαλώ εδώ στην έδρα ο κύριος Άρνολτ και μπορεί να μας μιλήσει για το θέμα του. Έχει έρθει ο κύριος Άρνολτ. Είναι παρόν ο κύριος Τόμ Άρνολτ, ο πρόεδρος ειδική ομάδας για την Ακροτική Αφρική. Θα καταφτάσει ανα πάσα στιγμή. Θέλει να προσθέσει κάτι η αντιπρόεδρος της ΔΕΒΕ, μήπως όσο αναμένουμε τον κύριο Άρνολτ.